Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε παρακαλώ την πρώτη μας ε, συνεδρίαση το 2018. Θα ήθελα να σε ευχηθώ καλή χρονιά, ευτυχισμένο το νέο έτος ε, σε όλους τους συναδέλφους, ε, τους συνεργάτες μας, του διερμηνείς, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστούμε και ανταποδίδουμε. Φαντάζομαι θα είναι δύσκολη χρονιά, πολύ άσχολη. Έχουμε πολλές ανακοινώσεις της Επιτροπής, ε, πολλές πολυμερείς διαπραγματεύσεις. Αλλά δεν είμαστε και άπειροι, είμαστε έμπειροι, ήδη είμαστε προς το τέλο τη θητεία, οπότε θα ανταπεξέλθουμε στα καθήκοντά μα σίγουρα. Επαναλαμβάνω και πάλι, καλή σα χρονιά. Και ξεκινάμε με μια μικρή καθυστέρηση της εργασίας της Επιτροπής Γεωργίας, αλλά πιστεύω ότι στην πορεία θα κερδίσουμε το χρόνο που χάσαμε κατά την έναρξη. Ε, σήμερα το πρόγραμμά μας είναι πλούσιο με πολύ σημαντικό, σημαντικά ζητήματα, με ε, καλεσμένος από την Επιτροπή Φυσικών Πόρων της Επιτροπής Περιφερειών αλλά και από την αντίστοιχη Επιτροπή της ε, Ευρωπαϊκής ε, Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής. Αυτά τα δύο όργανα είναι πολύ σημαντικά για μας, η Επιτροπή Περιφερειών και η ΕΟΚΕ. Και δεν έχουν μόνο συμβουλευτικό χαρακτήρα, αλλά και μεγάλη επιρροή τα δύο αυτά όργανα την διαμόρφωση των δικών μας συζητήσεων και των δικών μας ε, εργασιών. Και οι δύο επιτροπές ε, ε, περιφερειών και ΟΚΕ επηρεάζουν και η γνώμη τους έχει και βαρύτητα στις δικές μας εκθέσεις και γνωμοδοτήσεις. Και φυσικά ίδιοι είναι οι ψηφοφόροι γιατί είμαστε και στην Επιτροπή Περιφερειών και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αιρετοί. Ε, Επίση, στην Επιτροπή Περιφερειών έχουμε εκπροσώπους τη τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση, οπότε έχουν από πρώτο χέρι επαφέ με του ενδιαφερόμενου. Οπότε γι' αυτό είναι προ όφελό μα η στενή συνεργασία και σα ευχαριστώ θερμά για την ε, προθυμία σας να έρθετε και να μας παρουσιάσετε τις ε, ο Και ευχαριστώ και πάλι για την ε, στενή συνεργασία που έχουμε με τις δύο επιτροπές. Θα συζητήσουμε σήμερα λοιπόν ε, τα κοινά σημεία των γνωμοδοτήσεών μας. Αλλά αυτό αργότερα. Περνάμε στη κανονική σειρά των σημείων της σημερινής διάταξης. Έχουμε προσώπους σήμερα και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τους καλωσορίζω θερμά όλους και να ρωτήσω αν υπάρχουν παρατηρήσεις για την ημερήσια διάταξη. Αν όχι, να την εγκρίνουμε. Έχουμε διερμηνία από και προς 16 γλώσσες και επίσης ε, μεταδίδεται στο διαδίκτυο απευθεία η συνεδρίασή μας. Βάσει της διαδικασίας, θα ήθελα τώρα να εγκρίνουμε τα πρακτικά των προηγούμενων μας συνεδριάσεων της 13ης Νοεμβρίου, 22ης και 23ης Νοεμβρίου, 29ης Νοεμβρίου, 4ης Δεκεμβρίου, και 7 Δεκεμβρίου. Οπότε με τη γνωστή διαδικασία θα εγκρίνουμε τα πρακτικά. Περνάμε στο σημείο 4 τώρα της ημερήσιας διάταξης. Τα προβλήματα των νέων γεωργών. Μετά την μεταρρύθμιση της ΚΑΠ του 2013 ε, εξετάζουμε τις ε, πολιτικές ε, της εφαρμογής του προγράμματος στους νέους γεωργούς. Ο κύριος Καπούτο ανέλαβε την έκθεση για το σημείο αυτό. Θα θυμάστε ότι τον Οκτώβριο το τμήμα πολιτικής μας παρουσίασε 23 Νοεμβρίου το τμήμα πολιτικής μας παρουσίασε τη μελέτη για την εφαρμογή των πολιτικών των νέων γεωργών μετά την ε, μεταρρύθμιση της ΚΑΠ του 2013. Και μάλιστα διοργανώσαμε και δημόσια ακρόαση με το θέμα αυτό. Ε, τη σχετική έκθεση, όπως σας είπα, την ανέλαβε ο κύριος Καπούτο. Και μάλιστα η ακρόαση επικεντρώθηκε σε δύο θέματα. Την ε, ικανότητα της τρέχουσας ΚΑΠ και των μέτρων της να επιτύχει τους στόχους της ανανέωσης των γενναιών στη Γεωργία και τις προσδοκίες από την επόμενη ΚΑΠ που έχουν οι νέοι γεωργοί. Όλα αυτά τα συζητήσαμε γιατί γνωρίζουμε πόσο σημαντική είναι η νέη γεωργία για την Ευρωπαϊκή Γεωργία. Γνωρίζουμε ποια είναι η κατάσταση ό,τι αφορά την ανανέωση των γενεών στη γεωργία, που γίνεται σε πολύ χαμηλούς δυστυχώς ρυθμούς και αυτό μας δημιουργεί τεράστιες προκλήσεις. Μάλιστα, πολύ συχνά στην Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμού, στη συζήτηση της ε, έκθεσης ε, του ελεκτικού, του ελεκτικού συνεδρίου, είδαμε ότι για τους νέους γεωργούς υπάρχουν κάποια μέτρα ε, τη, της κοινή γεωργικής πολιτικής, αλλά δεν υλοποιούνται παρκώς και δημιουργείται ένα σημαντικό πρόβλημα. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε ποια είναι τα εισοδήματα των νέων γεωργών, αν είναι προσοδοφόρα η γεωργική απασχόληση και επίσης λόγω της ε, αυτοματοποίησης και της μηχανοποίησης η επιβάρυνση ε, είναι μεγάλη και δύσκολο είναι να ανταπεξέλθουν σε τέτοιες επιβαρύσεις και οικονομικές ε, οι νέοι Γεώργοι. Θα πρέπει λοιπόν να τονώσουμε την αγροτική ανάπτυξη και αυτό προϋποθέτει υποδομές και κοινωνικο-οικονομικές. Είναι πολύ διάστατο αυτό το πρόβλημα της βοήθειας των, προς τους νέους γεωργούς, αλλά αυτό το θέμα ίσως σε μερικές διαστάσεις ξεπερνά το εύρος της έκθεσης Καπούτο. Τώρα, επειδή έχουμε πολλά σημεία στην σε διάταξη, θα σας παρακαλούσα στο μέτρο του δυνατού να επιδείξω μία εγκράτεια στη χρήση του χρόνου αγόρευσης. Ακόμη και από τον εισηγητή ε, ζητώ κάτι τέτοιο. Α, ο κύριος Άγνιου, παρακαλώ. Και ποιο είναι το όριο του χρόνου αγόρευσης. Μπορούμε να βλέπουμε κάποιο χρονόμετρο γιατί είπατε να είμαστε λακωνικοί, αλλά πόσο λακωνικοί. Δώστε μας κάποιες ε, καθοδηγήσεις. Οι συντονιστές θα έχουν δύο λεπτά στη διάθεσή τους. Πρώτα όμως ο εισηγητής μας ο κύριος Καπούτο. Α, συγγνώμη, ο κύριος Δενανό. Όχι, όχι, για μετά, για τη συζήτηση. Για τη συζήτηση μετά ο κύριος Δενανό. Ο κύριος Καπούτο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Οπωσδήποτε θετικό ιονό το να ξεκινούμε το έτο συζητώντα για του νέου στη Γεωργία. Πολύ καλό ιονό για την Επιτροπή μα. 6% μόνο είναι αυτοί οι οποίοι διαχειρίζονται γεωργικέ εκμεταλλεύσει σε ηλικία κάτω των 35 ετών, ενώ το 50% έχει ήδη ξεπεράσει τα 50 χρόνια ηλικία στου γεωργού. Και αυτό είναι ένα γεγονός που πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη όταν συζητούμε την έκθεσή μου. Οι δύο αυτοί οι στόχοι λοιπόν που εξυπηρετούμε είναι και η ε, συλλογή και παροχή πληροφοριών σε σχέση με τα μέτρα τα οποία προβλέπονται στο πλαίσιο της κοινής πολιτικής για τους νέους και βέβαια έχουμε να κάνουμε μια πρώτη έκθεση αξιολόγηση της εφαρμογής σε επίπεδο Επιτροπής Γεωργίας ε, της οποίας εκθέσεως έχω και την τιμή να είμαι εγώ εισηγητής. Έχουμε λοιπόν στηριχθεί σε στοιχεία έρευνας της Επιτροπής Γεωργίας, ε, της έρευνας με τίτλο «Νέη Γεωργία επικαιροποίηση μετά την ε, μεταρρύθμιση του 2013 της κοινής γεωργικής πολιτικής», ε, έκθεσης που έχει, όπως ξέρετε, υποβληθεί στην Επιτροπή μας στις 23 Νοεμβρίου υπευλήθη στην Επιτροπή μας 23 Νοεμβρίου και ταυτόχρονα έχουμε και στοιχεία και από το ελεγκτικό συνέδριο και έχουμε διατυπώσει έτσι συστάσεις για τη βελτίωση του καθεστώτος που ισχύει για να ενισχυθούν οι γεωργοί νέα ηλικία να αντεπεξέλθουν στα μεγαλύτερα εμπόδια που αντιμετωπίσουν όσον αφορά την είσοδό του στον κλάδο της γεωργίας. Θα, θα αναπτύξω την παρουσίασή μου σε πέντε κύριους ε, κλάδους, για να κερδίσουμε και χρόνο βέβαια και θα αναφερθώ στη χρηματοδότηση όπου οπωσδήποτε θα χρειαστεί να βελτιωθεί το πρόγραμμα για τους νέους εισερχόμενους τους νέους γεωργούς και να ξεπεράσει το 2% σε εθνικό επίπεδο προκειμένου να ενθαρρύνονται οι νέοι να μπαίνουν στην γεωργία, να ενθαρρυνθεί δηλαδή η γενεαλογική ούτως ανανέωση. Τα πέντε χρόνια της ε, λειτουργίας της επιχείρησης αλλά και μια καλύτερη αντιμετώπιση των ε, επιτοκίων για τα δάνεια προς νέους γεωργούς χρειάζονται επανεξέταση, καλύτερη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, ε, Στρατηγικών Επενδύσεων, προκειμένου να εξασφαλιστούν λύσεις ικανοποιητικές για τους νέους γεωργούς σε όλα τα κράτη-μέλη. Το δεύτερο σημείο αφορά το ε, κρατικό, τη γραφειοκρατική επιβάρυνση, η οποία πολύ συχνά αποθαρρύνει τον νέο γεωργό, ενώ τα μέτρα θα έπρεπε να τον ενθαρρύνουν να ε, αναπτύξει μια γεωργική δραστηριότητα και εκμετάλλευση. Επίσης το συλλογικό ποσό της, των άμεσων επενδύσεων και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Γεωργικής Ανάπτυξης, Ανάπτυξη Πέθρου που θεωρούνται αρκετά περίπλοκο, ιδιαίτερα για τους νέους γεωργούς, οι οποίοι δεν έχουν εμπειρία προηγούμενη από τα συστήματα των πληρωμών. Το τρίτο θέμα έχει να κάνει με την πρόσβαση στη γη και την ε, αποδέσμευση των γεωργικών γεών, κάτι το οποίο χαρακτηρίζει το σκύριο εμπόδιο για τους νέους γεωργούς. Βεβαίως έχει να κάνει και με το σύστημα των άμεσων ενισχύσεων γιατί μια ελάχιστη αξιοποίηση της γης μπορεί να εξασφαλίσει σε κάποιον μακροπρόθεσμη εκμετάλλευση, δικαίωμα μακροπρόθεσμο εκμετάλλευση και διακράτηση της γης. Έτσι λοιπόν πρέπει να βρούμε λύσεις ε, που να εξασφαλίζουν και την πρόσβαση βέβαια στις επιδοτήσεις και την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των εδαφών μας προτείνω την ενίσχυση των απαραίτητων για την χορήγηση των επιδοτήσεων δραστηριοτήτων, την αύξηση του ποσοστού δραστηριότητας, έτσι ώστε να ε, υπάρχει αυτό και ταυτόχρονα να συνδέεται η χορήγηση επιδότησης με την ανάπτυξη συγκεκριμένων κοινωνικού χαρακτήρα ή περιβαλλοντικού χαρακτήρα αγαθών μέσα από τη γεωργική ε, αξιοποίηση, γεωργική εκμετάλλευση. Επίσης θα πρέπει να συμβάλλουμε στην κινητικότητα των ε, γεών και ζητούμε μια νομοθετική πρόταση που θα ενισχύσει την εγκαθίδρυση εθνικών προγραμμάτων που θα προωθούν την ε, κινητικότητα των γεών και την διαδοχή στις, ε, στην εκμετάλλευση των γεών. Έτσι θα υπάρχουν ενδεχομένως κίνητρα για τον πιο ηλικιωμένο γεωργό να μεταφέρει τη γη του, ε, κληροδοτεί τη γη του σε νεότερους ή να εκχωρεί τη γη του σε νεότερους γεωργούς. Αυτό μέσα και από συστήματα ενδεχομένω προόριστα ταξιοδότηση. και ταυτόχρονα θα, θα πρέπει να ενισχυθούν και να ενθαρρυνθούν μέσω των εταιρικών σχέσεων, μακροπρόθεσμης, χρονομίστοσης αλλά και άλλων ε, ταμείων που θα μπορούσαν να οργανωθούν σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο οι νέοι γεωργοί ώστε να διευκολύνονται και να υπάρχει και μια επικοινωνία μέσα από τις υπηρεσίες ε, φερρυπίν ε, κινητικότητα των γεών που θα επιτρέπει την επικοινωνία μεταξύ νέων και πιο ηλικιωμένων γεωργών για να ε, διευκολυνθεί αυτή η διαδοχή. Υπάρχουν δραστηριότητες που χρειάζεται οπωσδήποτε και να εξεχρονιστούν και να χρηματοδοτηθούν με καλύτερα πιο ικανοποιητικά από τον προπολογισμό και δηλαδή τον ευρωπαϊκό. Ταυτόχρονα και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν περισσότερε δυνατότητε κατάρτιση για νέου νέους που ενδιαφέρονται να γίνουν γεωργοί, αλλά και για ε, γεωργούς που ήδη έχουν αναπτύξει την ε, δραστηριότητά τους. Θα πρέπει να ενισχυθεί η επικοινωνία, η χρηματοοικονομική συνεργασία, η καινοτομία ασφαλώς και ε, κέριο σημείο για την ανάπτυξη της γεωργικής μας οικονομίας με νέες δραστηριότητες, καινοτόμες και σύγχρονες δραστηριότητες, ώστε να καταστεί και πιο ενδιαφέρουσα, πιο ελκυστική για τον νέο η Γεωργία. Πρέπει να ενισχύονται και οι ψηφιακές και καινοτόμες γεωργικές δραστηριότητες και καλό την Επιτροπή μας αυτό να καταγράφεται σε κάθε μελλοντική ε, μεταρρύθμιση της ΚΑΠ. Αυτά είναι τα κέρια σημεία, αυτά είναι τα κεντρικά σημεία της εκθεσεώς μου, που βεβαίως έχει σημασία πολύ μεγάλη και κεντρική να προωθηθεί από όλες τις πολιτικές ομάδες, να στηριχθεί από όλες τις πολιτικές ομάδες. Με αυτό το πνεύμα λοιπόν διατυπώνω και την απόλυτη διάθεσή μου προς συνεργασία. Η προθεσμία για την κατάθεση των τροπολογιών, υπενθυμίζω στους συναδέλφους, έχει προσδιοριστεί για τις 19 Ιανουαρίου. Η ψηφοφορία στην Επιτροπή μας προβλέπεται για τις 23 Απριλίου. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Καπούτο. Θα ήθελα να προσθέσω ότι ε, δύο λεπτά δικαιούνται και οι σκιώδεις συγκητές που παρακολουθούν ε, τη διαμόρφωση των εκθέσεων. Ο πρώτος σκιώδης συγκητής είναι ο κύριος Γιάνν Χόιτεμα, Παρακαλώ. Δύο λεπτά κι εσείς. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την εξαιρετική του έκθεση. Κατέβαλε σημαντικέ προσπάθειε και, και νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή βάση για περαιτέρω συζητήσει. Επεσήμανε πέντε σημεία με πολύ καλά δομημένο τρόπο που μου άρεσε ιδιαίτερω. Εν γέννη, θεωρώ ότι θα πρέπει να δούμε πώ μπορούμε όντω να προσελκύσουμε ε, τους ε, νέου γεωργού και είναι πολύ σημαντικό να επικεντρωθούμε στην καινοτομία, να εξετάσουμε και τις ε, προκλήσεις του μέλλοντος ε, και μου άρεσε πολύ που το συμπεριέλαβε αυτό στην έκθεσή του. Μετά κατάρτιση και άλλα ζητήματα που μας επιτρέπουν να ε, συνδυάσουμε τις επιμέρους γενιές για να υπάρξει έτσι μια σωστή διαδοχή. Αυτό είναι ενδιαφέρον για το διοικητικό άχθος. είναι σωστές οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να έχουμε μία προσέγγιση προσανατολισμένη προς τα αποτελέσματα. Νομίζω ότι αυτό είναι κρίσιμη σημασία για τις νέες γενιές. Έχουν πολλές νέες ιδέες και νομίζω ότι με μια νέα τέτοια προσέγγιση μπορούμε να αφήσουμε τον απαραίτητο χώρο να αναπτυχθούν αυτές οι νέες ιδέες και να αφήσουμε τους νέους να το κάνουν μόνοι τους, να δουν πώς θέλουν να πετύχουν τους στόχους ε, που θέτουμε εμείς στην Ευρώπη για την βιωσιμότητα, το περιβάλλον, αντί να επιβάλλει κάποια μέτρα, να επιβάλλουν οι Βρυξέλλες κάποια μέτρα και να τους ε, λέμε τι πρέπει να κάνουν, να βρουν μόνο τους τον δρόμο. Μετά για την ε, υφιστάμενη κοινή πολιτική και την πρόσβαση στις γεωργικές εκτάσεις θα πρέπει να δούμε με μεγάλη προσοχή τις αρνητικές επιπτώσεις ε, που ενδεχομένως να υπάρχουν έστω και άθελά μας της κοινή γεωργικής πολιτικής που μπορεί να έτσι να οδηγεί σε αύξηση των τιμών της γης ή των ε, συμβάσεων μισθώσεων και αυτό ε, δυσχεραίνει την μεταφορά της γης στη νεότερη γενιά. Πρέπει να εξετάσουμε με προσοχή λοιπόν την κοινή γεωργική πολιτική για τυχόν τέτοιες αρνητικές επιπτώσεις. Ευχαριστώ. Μάλιστα, παίρνουμε στους υπόλοιπους ομιλητές 1,5 λεπτό, γιατί είναι σημαντικό το θέμα και έχουμε θέμα αρκετό για συζήτηση. Ο κύριος Ντενανό, 1,5 λεπτό. Ντενανό, 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πράγματι, η έκθεση είναι εξαιρετικά σημαντική που θα προσδιορίσει το μέλλον της Γεωργίας στην Ευρώπη και θα ήθελα ε, να σταθώ ακριβώ σε αυτά τα στοιχεία, γιατί η δυσκολία για τους νέους είναι η πρόσβαση στη γη. Συχνά η πρόσβαση στη γη είναι κάτι το οποίο δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να αποκτήσουν ε, οι γεωργοί. Ε, κάποιοι βέβαια σαν οικογενειακό πλαίσιο μπορούν ε, να λάβουν τη γη μέσω κληρονομιά. κάποιοι από τους συγγενείς του Οι υπόλοιποι όμω πρέπει να αγοράσουν τη γη. Πρέπει λοιπόν να να βρούμε άλλους ε, τρόπους ε, ε, χρήσης της γης πέραν της άμεσης απόκτησης και αγοράς. Υπάρχουν λοιπόν άλλες τέτοιες μέθοδοι που επιτρέπουν ακριβώς την εγκαθίδρυση και την εγκατάσταση αυτών των γεωργών και τη χρήση της γης. Μετά υπάρχει και μία σπατάλη γης ε, Στι αστικοποιημένε ζώνες θα πρέπει να ε, δώσουμε μεγάλη προσοχή για να μην εγκαταλείπουμε τη γεωργία ε, για να οικοδομούμε μονοκτήρια. Πρέπει να υπάρχει ισορροπία σε αυτό το επίπεδο και οι εθνικοί νόμοι να προστατεύουν τη γεωργία και σε αυτές τις ζώνες που είναι ιδιαίτερα ευάλωτες, γιατί είναι πολύ ε, χρήσιμες ε, για τη Γεωργία και έτσι θα πρέπει να δώσουμε μεγάλη προσοχή σε αυτό το ζήτημα. Άλλο ζήτημα που τίθεται είναι αυτό των υποδομών. Όταν, ε, για παράδειγμα, οικοδομούμε είτε έναν αυτοκινητόδρομο, είτε έχουμε έργα υποδομών για ένα αεροδρόμιο, πρέπει με μεγάλη προσοχή να εξετάσουμε ε, για να αποφύγουμε τον ε, καταγερματισμό ε, της γης και έτσι να μπορέσουμε να προσελκύσουμε και γεωργούς. Πρέπει να προτείνουμε επίσης ένα διαφορετικό ε, τρόπο ε, και μέθοδο, μια διαφορετική μέθοδο καλλιέργειας πιο παραδοσιακή. Συμπαθάτε με που θα κάνω ένα σχόλιο τώρα, αλλά στην πατρίδα μου έχουμε αγροτεμάχια που έχουν μετατραπεί σε οικόπεδα και μπορούν να στεγάσουν 150 εκατομμύρια ανθρώπους. Ε, γιατί μερικές φορές θέλουμε να εξασφαλίσουμε τη ροή των κεφαλαίων προς την, ε, προς την Ήπεθρο. Ε, 150 εκατομμύρια όντως, μπορεί να στεγάσουν 150 εκατομμύρια ανθρώπους. Ε, είναι σημαντικό πρόβλημα αυτή η αξιοποίηση των αγροτεμαχίων για οικιστικούς λόγους. Ο κύριος Σάντος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όντως η Γεωργία και οι νέοι αγρότες στη Γεωργία αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα όπως ακούσαμε. Και όπως είπε και ο Νικολά Καπούτο, ε, γυράσκει και ο γεωργικός πληθυσμός. Γι' αυτό θα πρέπει να βρούμε τρόπους για να ενισχύσουμε την ηλικιακή ανανέωση. Το 60% των γεωργών ε, είναι άνω των 65 ε, ετών. είναι ελάχιστο το ποσοστό των ε, νέων αγροτών. Είναι σημαντικό λοιπόν να δώσουμε έμφαση στην ηλικιακή ανανέωση στη γεωργία. Είναι κρίσιμο σημείο, νευραλγικό. Είναι αδιανόητο ένα ε, γεωργικό κόσμο χωρί γεωργού. Θα πρέπει λοιπόν να καταστήσουμε προσοδοφόρα αυτή τη γεωργική δραστηριότητα για να προσελκύσει του νέου. Υπό την επιφύλαξη των κοινωνικο-οικονομικών φαινομένων που μπορεί να οδηγούν σε μια αντίστροφη τάση. Έγιναν κάποιες, ε, κάποιοι πρόοδοι στον κανονισμό Omnibus και ε, συμφωνούμε και με τις προτάσεις του κυρίου Καπούτο. Θα πρέπει να εξοικειωθούν οι νέοι με τις γραφειοκρατικές διαδικασίες για την πρώτη κατάσταση. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε κίνητρα για τη μεταβίβαση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και να ενισχύσουμε την θετική διάκριση υπέρ των νέων αγροτών. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, κύριος Μπόγκοβιτς. <clears throat> E, zelo pomembno področje. E, podpiram to, kar je zapisano. Ευχαριστώ πολύ και υποστηρίζω την ε, έκθεση και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων, ιδιαίτερα για τους ε, νεαρούς γεωργούς, ε, όπως προτείνεται στην έκθεση και μάλιστα θεωρώ πολύ πρόσδεκτο και το μέτρο της ε, πρόορης ταξιοδότησης Υπάρχουν διάφορα μέτρα στην ε, πρόταση Omnibus, αλλά χρειάζονται ακόμη περισσότερα για να εξασφαλίσουμε ένα θετικό μέλλον, ένα καλό μέλλον για τους νέους μας, γιατί θα μείνουν στην Ήπεθρο, στη γεωργική δραστηριότητα, μόνο αν έχουν ένα καλό εισόδημα και καλό επίπεδο ζωής. Ε, ε πρέπει λοιπόν για να το καταφέρουμε αυτό ε, να γνωρίζουμε ότι θα υπάρχουν λιγότερες διαθέσιμε θέσεις εργασίας στη Γεωργία γιατί θα είναι και λιγότερη διαθέσιμη γη. Άρα θα πρέπει να επιδιώξουμε την διαφοροποίηση, την επαγγελματική στις εκμεταλλεύσεις. Θα χρειαστούμε υποδομές περισσότερες, διαδίκτυο και διαφοροποίηση και δραστηριοτήτων, ε, διαφορετικές ε, δραστηριότητες, φερρυπίν, ε, παραγωγή τυριού, τουριστικές δραστηριότητες, κοινωνικές υπηρεσίες επίσης που είναι πολύ σημαντικές για την Ήπεθρο αλλά πρέπει να εξασφαλίσουμε και κινητικότητα και καλύτερες ενεργειακές δομές. Όλα αυτά έχουν ξεκινήσει σε προπαρασκευαστική φάση με προγράμματα εφιών χωριών. Θα τα συζητήσουμε στον Μπλέτ τον Απρίλιο. Με, την, με τους επιτρόπους Μπούρτς και Χόγκαν που θα έρθουν στην διάσκεψη αυτή, με την ελπίδα πάντα ότι θα μπορέσουμε και να προσελκύσουμε και άλλα χρήματα πέραν του, και του Γεωργικού Ταμείου, αλλά και κοινωνικά και άλλα ταμεία. Η κυρία Πετήρ τώρα. Όταν βλέπετε ότι σηκώνω το σφυράκι, ε, να έχετε υπόψη ότι πλησιάζετε προς το τέλος του χρόνου, γιατί δεν είναι εύκολο να κοιτάει κανείς πάντα το χρονόμετρο. Αλλά κοιτάξτε όταν σηκώνω το σφυράκι. Η κυρία Πετήρ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και συγχαίρω τον κύριο Καπούτο για την πολύ αξιόλογη έκθεσή του. Πραγματικά είναι άρτια και θα ήθελα να συμβάλλω και εγώ με μερικές προτάσεις. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό να δώσουμε κίνητρα και να στηρίξουμε ε, την ε, διαδοχή των γενεών και τη μεταβίβαση των γεών, γιατί σε πολλές περιπτώσεις πολύ αργά γίνεται η μεταβίβαση από πιο ηλικιωμένους σε νεαρότερους γεωργούς. Θα πρέπει να δώσουμε κίνητρα στους νέους αγρότες για να ασχοληθούν με τη γεωργία. Επίσης, ε, θα πρέπει ε, να λάβουμε υπόψη και τους ηλικιωμένους. Στην ε, ε, Κροατία σχεδόν όλοι οι συνταξιούχοι που ήταν προηγουμένω γεωργοί έχουν πενιχρές συντάξεις, άθλιες κάτω από το κατόφλι της φτώχειας. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε ελάχιστα όρια κρατικών ε, συντάξεων ώστε να μην αναγκάσουμε τους γεωργούς τους στη ζωή σύτιζαν ε, εμάς να χρειάζεται να περάσουν ε, μία ε, τρίτη ηλικία πεινώντας. Επίση θα πρέπει να εξετάσουμε το θέμα των επιτοκίων στην Κροατία. 8% είναι το επιτόκιο για τους αγρότες, ενώ σε άλλες χώρες είναι 0,2% είναι αδύνατο να αντέξουν τόσο υψηλά επιτόκια. Είναι και αδύνατο να είναι ανταγωνιστικοί με τόσο υψηλά επιτόκια οι Κροάτες αγρότες. Επίσης, σε ό,τι αφορά την πενταετή περίοδο ε, για την διάρκεια που μπορούν να αξιοποιήσουν αυτές τις επιχορηγήσεις, συμφωνώ με το μέτρο που πρότεινε το ελεκτικό συνέδριο. Θα πρέπει επίσης να γίνει διάκριση μεταξύ των νέων αγροτών και των ε, πρωτοεισερχόμενων στη Γεωργία, που δεν είναι κατά ανάγκη και νέοι. Ευχαριστώ κύριος Αντριέ. Euh, Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ πλευρά μου να ευχαριστήσω τον κύριο Καπούτο για την ποιότητα ε, της έκθεσής του. Τέσσερις ε, παρατηρήσεις από πλευρά μου. σε ό,τι αφορά την ε, πρόσβαση στις επιδοτήσεις. Σε ό,τι αφορά το κληρότημα προς νέους αγιοργούς, είναι ένα βασικό εργαλείο για την ε, εγκαταστασή τους. Δεν είναι υποχρεωτικό σε όλα τα κράτη-μέλη και θεωρώ ότι θα πρέπει να γίνει αυτό το μέσο υποχρεωτικό ε, και να προσαρμόσουμε τις τους όρους ε, πρόσβαση. Συμφωνώ με την κυρία Πετήρ για τόσο είπε για τη δεξιοδότηση γιατί είναι κάτι που πρέπει να συνδεθεί, να το συνδέσουμε εδώ και το μέτρο της πρόορης δεξιοδότηση ε, είναι ένα καλό εμέσο αρκεί να συνδέεται και με την... Διακόπτεται. Διακόπτει ο Πρόεδρος, υπάρχει πρόβλημα με την αγγλική διερμηνία. Παρακαλώ αφαιρέστε όμω ε, την ε, παρέμβαση του συναδέλφου από τον χρόνο μου. Συνεχίζω λοιπόν. Δεύτερον, ενεργός γεωργό. είναι κάτι το οποίο ανέφερε και ο εισηγητή και θα πρέπει να εξετάσουμε αυτό το ζήτημα για να δώσουμε πρόσβαση ε, στα εργαλεία χρηματοδότηση τη κοινής γεωργικής πολιτικής. Θα είναι μια συγκεκριμένη τροπολογία αυτή. Ε, πρέπει όμως να υπάρχει ενδεχομένως και ένα πλαφόν. Είναι ζητήματα τα οποία θα εξετάσει η μελλοντική μεταρρύθμιση, όμως θα πρέπει να το εξετάσουμε. Και τέλος, πρέπει ε, να ενισχύσουμε ε, την ασφάλιση της γεωργίας που θα είναι κεντρικό σημείο στην μελλοντική κοινή γεωργική πολιτική γιατί υπήρξε σημαντική απορρίθμιση και απελευθέρωση της οικονομίας. Ε, πρέπει λοιπόν, είναι κρίσιμη σημασία να ε, επανεξετάσουμε την κοινή γεωργική πολιτική για να διασφαλίσουμε και το μέλλον της γεωργίας και και το ζήτημα της περιβαλλοντικής καινοτομία, αλλά και το θέμα της κινητικότητας των γεωργών. Είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να ε, δίνουμε κίνητρα για την ε, κινητικότητα προκειμένου να υπάρχει ανταλλαγή βέλτιση πρακτικών μεταξύ χωρών, μεταξύ περιφερειών και έτσι να θεσπίσουμε ένα πραγματικό δίκτυο. Κύριο Βάιτς, Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Λαμβάνω το λόγο εκ προσωπώντας την κυρία Χόιμπουχ, τη σκιώδη συγγητριά μας, ευχαριστώντας καταρχάς τον κύριο Καπούτο για την εξαίρετη έκθεση, ένα-δύο σημεία θέλουμε να ε, τονίσουμε ιδιαίτερα για, τους νέους, ε, για μια διαφοροποίηση μεταξύ νέων γεωργών και νέων εισερχόμενων στη γεωργική δραστηριότητα γιατί εκεί ε, είναι πολύ σημαντικό να τους υποστηρίξουμε τους νέους εισερχόμενους ακόμα και όταν είναι άνω των 40 ετών ηλικίας. Επίσης πρέπει να προσφέρουμε, να τονίσουμε περισσότερο το θέμα της κοινωνικής ή περιβαλλοντικής συνεισφοράς της γεωργίας, περιορισμό των κλιματικών συνεπειών ή αλλαγών, ενίσχυση ενίσχυση της ε, γονιμότητας της γης, ε, κτηνοτροφία κτλ. Όλα αυτά πρέπει να προωθούνται και να τονίζονται ιδιαίτερα. Σημαντικό επίσης είναι το θέμα της πρόσβασης στις γεωργικές γης και εδώ θα πρέπει και μπορεί νομίζω η ΚΑΠ να ε, εισαγάγει πολλά ακόμη μέτρα στοχευμένα επιδοτούμενα δάνεια, φερρυπίν, δάνεια με επιδοτούμενο επιτόκιο δηλαδή, ε, αναδιανομή γης με τρόπο ώστε να επιτρέπεται η πρόσβαση και σε μικρότερες εκμεταλλεύσεις στη γη, περιορισμό της αναλογίας της επιδότησης ως προς το εκτάριο ώστε να μην ευνοούνται οι μεγάλες εκμεταλλεύσεις και γενικότερα διευκόλυνση για τον νέο και νεοεσερχόμενο γεωργό της πρόσβασης στη γη. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ροπέ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, θεωρώ το θέμα αυτό πολύ σημαντικό και είναι ενδεικτικό ότι με αυτό το τόσο σημαντικό θέμα ξεκινάμε τη νέα χρονιά. Και ευχαριστώ τον εισηγητή και όσους συνέβαλαν στην διαμόρφωση αυτού του εγγράφου. Ήρθε επιτέλους η ώρα να ασχοληθούμε με το ζήτημα αυτό. Τώρα που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει την πρόταση των νέων δημοσιονομικών προοπτικών. Οπότε θα πρέπει να εξετάσουμε ε, το πώς θα συμπεριλάβουμε όλες αυτές τις σημαντικές πτυχές στο νέο δημοσιονομικό πλαίσιο και πώς θα ε, συνεκτιμήσουμε και την προοπτική του νέου αγρότη στο έγγραφο αυτό. Ό,τι κάνουμε σήμερα θα επηρεάσει το μέλλον μας, το σύστημα μετά το 2020. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις εξελίξεις στη Γεωργία. Γνωρίζουμε την κατάσταση για τους νέους αγρότες. Θα πρέπει όλα αυτά να τα περιλάβουμε στα κείμενά μας. Μόνο έτσι θα αλλάξουμε την κατάσταση και θα βελτιώσουμε το μέλλον. Για να μην μείνουμε μόνο στα λόγια και να περάσουμε και στα έργα. Ε, θα πρέπει να δούμε το εισοδηματικό χάσμα που υπάρχει μεταξύ του παραγωγικού κλάδου και της βιομηχανίας. Η διαφορά ε, βρίσκεται στο 50 με 60%. Τόσο είναι το ε, οικονομικό κενό. Και μάλιστα στην Ευρώπη η Γεωργία είναι μορφωμένη. Ε, μάλιστα οι νέοι σπουδάζουν, οπότε γιατί να διαλέξουν τη γεωργία αν δεν είναι προσοδοφόρος αυτή η γεωργική δραστηριότητα. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε κίνητρα λοιπόν για να προσελκύσουμε τους νέου στη γεωργία. Επίση, όσοι κληρονομούν την αγροτική εκμετάλλευση είναι σε πολύ ευνοϊκότερη κατάσταση. Ενώ για του άλλου που δεν έχουν ε, μια τέτοια κληρονομιά είναι δύσκολο ε, να έχουν μια πρόσβαση σε γεωργική εκμετάλλευση. Ο κύριο Άγνιου. Ευχαριστώ. Σημαντική έκθεση επικρίνει τον τρόπο με τον οποίο ε, ο πρώτος πυλώνος ουσιαστικά επιβραβεύει την ε, κτήση ιδιοκτησία γης. Ε, στηρίζω λοιπόν αυτό που αναφέρεται, όμως θέλουμε εδώ να επιβάλλουμε πιέσεις προς τα κράτη-μέλη για να αλλάξουν τις νομοθεσίες τους. Όμως αυτό να πω στα κράτη-μέλη. Και στο παρελθόν έχω προτείνει να υπάρχει ε, ο μηχανισμό συνταξιοδότηση ε, των γεωργών, που η σύνταξη να είναι πολλαπλάσια των προηγούμενων επιδοτήσεων που έχει λάβει, επί 5 για παράδειγμα. Ε, αυτό μετά δεν θα μπορεί πλέον να πάρει επιδοτήσεις και έτσι θα υποτιμάται και η αξία του αγροταμαχίου, ίσως να μπορεί μετά και ένα νέο γεωργό να το αποκτήσει. Πολύ συχνά υπερβαίνουμε εδώ ε, τα δημοσιονομικά περιθώρια. Πρέπει λοιπόν να ε, είμαστε προσεκτικοί. Πάντα θα πρέπει να υπάρχει κατάρτιση για οποιονδήποτε μπαίνει στην γεωργία. Αν η αξιολόγηση γίνεται μόνο με συγκεκριμένα παιδεία, με ένα συγκεκριμένο checklist, ε, το εξετάζουμε μόνο ως επάγγελμα, αλλά είναι κάτι παραπάνω από ένα απλό επάγγελμα. αυτοί που είναι σε καλύτερη θέση να αξιολογήσουν αν μπορούμε να δανείσουμε χρήματα σε έναν νέο γεωργό είναι οι τοπικές τράπεζε. Και θα ήθελα να εξετάσω, να δω μάλλον ε, τα ε, δημόσια αυτά κονδύλια να χρησιμοποιούνται ως ε, εγγύηση αυτού του δανείου. Γιατί δεν έχουν τα περιουσιακά στοιχεία αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι νέοι, για να αποκτήσουν ένα δάνειο. Και αν μπορούμε έτσι αν μπορεί η κυβέρνηση να σταθεί εγγυητή, για παράδειγμα, αυτό θα ήταν ε, πολύ ωφέλιμο. Υπάρχουν και άλλες ε, μέθοδοι ε, κοινή ε, χρήσης της γης, όπως υπάρχει και στη Νέα Ζηλανδία. Τέλος, πρέπει να έχουμε καλύτερη και πιο απλή νομοθεσία. Είναι κάτι το οποίο θα μας βοηθούσε. Κυρία Γκαρσία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ με τους προλαλήσαντες ότι η έκθεση μας είναι πολύ σημαντική και ευχαριστώ τον εισηγητή μας τον κύριο Καπούτο για την πολύ αξιόλογη προσπάθειά του. Ε, συμφωνώ με πολλές προτάσεις του εισηγητού, αλλά άλλες προτάσεις του με προβληματίζουν. Για παράδειγμα, λέει ότι όντω ε, συμφωνώ ότι υπάρχουν προβλήματα με τη γεωκτησία. Όταν λέτε όμω ότι θα πρέπει να αυξηθεί το επίπεδο δραστηριοτήτων ώστε να δικαιούται κάποιο ε, ενισχύσει, αυτό ίσω οδηγήσει μια βεβαιότητα στον κλάδο ε, αρνητική. Δηλαδή αβεβαιότητα. Γι' αυτό θα ήμουν πολύ επιφυλακτική ως προς την πρότασή σας αυτή. Επίσης, μετά την τελευταία αναθεώρηση της ΚΑΠ με τον κανονισμό Omnibus, έχουμε την τύχη να έχουμε πια νέα μέτρα και αύξηση και βελτίωση της ε, πληρωμής ενισχύσεων στους νέους αγρότες. Να δούμε λοιπόν πώς θα εφαρμοστούν αυτά τα νέα μέτρα του κανονισμού Omnibus στην κοινή γεωργική πολιτική πριν προτείνουμε εμείς νέα μέτρα. Είναι αλήθεια ότι ένας από τους πιο σημαντικούς στόχους της κοινής γεωργικής πολιτικής με βάση ε, την ανακοίνωση του κυρίου Χόγκαν που δημοσιεύθηκε στις 29 Νοεμβρίου, ε, το πιο σημαντικό θέμα που εντοπίζει ο Επίτροπος είναι η ηλικιακή ανανέωση και θα πρέπει να γίνουν οικονομικές προσπάθειες για να υποστηριχθεί αυτή η ανανέωση των γενεών, η ηλικιακή ανανέωση. Επίσης, ε, έχουμε ένα πολύ στενό χρηματοδοτικό πλαίσιο στην κοινή γεωρική πολιτική. Προσοχή λοιπόν, α μην προτείνουμε από τώρα πρόσθετα μέτρα και να μην βάλουμε όλη την οικονομική μας προσπάθεια στο ίδιο καλάθι. Να έχουμε μια διαφοροποίηση των μέτρων. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος. Εμείς στην Επιτροπή Γεωργίας να μην γουρσουζεύουμε ότι θα γίνει οπωσδήποτε περιορισμός του γεωργικού προϋπολογισμού. Ας μην τα λέμε εμείς αυτά. Ο κύριος Νέκοφ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα κύριε Πρόεδρε να ευχαριστήσω τον Νικόλα Καπούτο για την ε, πολύ αξιόλογη αόρτη έκθεσή του. Να συμφωνήσω πλήρως με τη στάση του και κυρίως την σύσταση να αυξηθεί το μέγιστο επίπεδο χρηματοδότησης πάνω το 2% και επίσης να βελτιώσουμε την πρόσβαση στη γη για τους νέους αγρότες. Αυτή είναι η σημαντική πρόκληση γιατί η ιδιοκτησία έχει γίνει στόχος των κερδοσκόπων ε, και είναι όλο και πιο δύσκολη η πρόσβαση των γεωργών στη γη. Επίσης, οι νέοι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλούς περιορισμούς, ιδιαίτερα στις ορεινές περιοχές και τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των ορεινών περιοχών είναι ακόμη πιο προβληματικά. Και μάλιστα η γεωργία είναι από τις ελάχιστες δυνατότητες ε, οικονομικής ε, δραστηριότητας που έχει ο πληθυσμός εκεί. Θα πρέπει λοιπόν να ληφθούν υπόψη οι και των ε, επιμέρους περιοχών. Θέλουμε ένα στοχευμένο ε, πρόγραμμα στήριξης για τους νέους αγρότες, ιδιαίτερα στις ορεινές περιοχές. Θα μπορούμε να έχουμε ένα συντελεστή, πολλαπλασιαστή, για να λαμβάνει υπόψη και τη διάσταση της γεωργίας, αλλά σε ορεινές συνθήκες. Ε, να λαμβάνουμε υπόψη τις αρρώσιμες καλλιέργειες, ε, την εσοδεία, το επίπεδο της κτηνοτροφίας και όλα αυτά να ληφθούν υπόψη σε ένα συντελεστή για να στηρίξουμε περισσότερο τους παραγωγούς που ε, δραστηριοποιούνται σε δύσκολες συνθήκες όπως είναι στις ορεινές περιοχές. Γιατί παραλαμβάνω έτσι θα συμβάλλουμε στην δημιουργία και στην διαφύλαξη γεωρικών δραστηριοτήτων και στις αντίξουες συνθήκες των ορεινών περιοχών. Έχω και άλλες προτάσεις, έτσι τις υποβάλλω γραπτός. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Ε, Κύριο Φλάνναγκαν, πολύ ενδιαφέρουσα και σημαντική έκθεση. Το πιο σημαντικό όμω από όλα, και νομίζω ότι είναι και το πιο σημαντικό για οποιονδήποτε, σε οποιαδήποτε δραστηριότητα επαγγελματική και αν είναι, είναι να μπορεί να βγάλει τον βιοπορισμό του εάν δεν έχει κέρδο ο γεωργό ή ο νέο ο οποίος ενδιαφερόταν ενδεχομένω για τη γεωργία δεν πρόκειται να μπει στο γεωργικό επάγγελμα. Αυτό λοιπόν είναι το κύριο κριτήριο και έχουμε σχετικά καλές προτάσεις σε σχέση με την πρόταση Omnibus που οφείλουμε βέβαια στου συνεισηγητέ. αλλά πάλι παραμένει το φαινόμενο ένα γεωργό να έχει ε, να αποκλείεται πλήρως από το πλαίσιο της ενίσχυσης εάν έχει για πενταετία και άνω ή μη απασχόληση ή μερικού χρόνου μόνο απασχόληση. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να μας επιτρέψει να συνεχίσουμε. Δεν υπάρχουν επαρκή χρήματα για το νέο γεωργό. Εάν θέλει κάποιο να μπει δηλαδή στη γεωργική δραστηριότητα μπορεί να διατηρεί κάποιο άλλο στη γη χωρίς να κάνει τίποτα ουσιαστικά. Βεβαίω και χρειάζονται υπηρεσίε οι νέοι όπω και οι πιο ηλικιωμένοι. Φερρυπίν, εάν κάποιο πάθει ένα ατύχημα στη χώρα μου λόγω της λιτότητας και λόγω του ότι είμαστε υποχρεωμένοι να ξεπληρώνουμε τα, τραπεζικά, τα χρέη μάλλον των τραπεζών δεν έχουμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε υγειονομικές υπηρεσίες, υπηρεσίες υγείας στην Ήπεθρο σε κάποιον ο οποίος ενδεχομένως να έχει πάθει έμφραγμα. Μπορεί να μείνει στον τόπο και να μην φτάσει στο νοσοκομείο. Χρειάζονται σχολεία, χρειάζονται ε, υπηρεσίες ε, ευρυζωνίας. Ε, όλα αυτά λοιπόν για να μπορέσει να επιβιώσει η Πεθρός και όλα αυτά για να στηρίξουμε και τη δυνατότητα του πιο ηλικιωμένου γεωργού να βγει στη σύνταξη και να ανοίξει το δρόμο για τους νεότερους γεωργούς. Όλα αυτά πρέπει να τα διευκολύνουμε. Και βεβαίως το κύριο είναι να είναι επικερδής δραστηριότητα η γεωργική δραστηριότητα. Γιατί να κάτσει ο γεωργός όλο το χρόνο να αγωνίζεται αν δεν μπορεί να εξασφαλίσει τα προστοζήν. Και κάτι ακόμη για, τους για τον πρόεδρο και το χρόνο που δίδεται στους ομιλητές και τους ηγητές. Είπατε αρχικά δύο λεπτά ε, γιατί είναι σημαντικό να είμαστε οικονόμοι στο χρόνο. Μετά έγινα 1,5 λεπτό. Δεν κατάλαβα γιατί ξαφνικά έγινε λιγότερο σημαντική η δική μου η παρέμβαση από τον προλαλισάντων. Κατά 30 μάλιστα δευτερόλεπτα. Δεν είναι δίκαιο αυτό, Πρόεδρε. Δίκαια έχετε κύριε Φλάναγκαν. Όταν ε, προχωρεί ο χρόνος αρχίζω και κουνάω το σφυράκι. Για να σε πιστήσω την προσοχή ότι πλησιάζεται προς το τέλος του χρόνου. Κύριε Βούδα, χρόνια πολλά γιατί έχετε και γενέθλια σήμερα αν δεν κάνω λάθος. Ευχαριστώ. Χαιρετίζω την έκθεση του κύριου Καπούτο στη χώρα μου έχει οδηγήσει ορισμένε συζητήσει που αφορούν το γεγονό ότι όσοι συνταξιδοτούνται και λαμβάνουν έτσι σύνταξη από το κράτο, εξαιρούνται και αποκλείονται από ε, τι επιδοτήσει. Δεν μπορούμε να δεχθούμε αυτή την προσέγγιση, γιατί και οι συνταξιούχοι, από όπου και απένουν σύνταξη, θα πρέπει να έχουν ε, ίση πρόσβαση στι επιδοτήσει γιατί πολύ συχνά οι συντάξει είναι χαμηλέ, ιδίω ε, στι χώρε της Ανατολική Ευρώπη. Σε ό,τι αφορά τώρα τη συγκέντρωση γη, αυτό είναι ένα υπαρκτό πρόβλημα, ιδίω στη Ρουμανία. Και εδώ θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, γιατί αυτό το φαινόμενο περιορίζει την πρόσβαση των νέων στη γη και των νέων γεωργών στη γη. και μάλιστα επικεφαλής αυτής της προσπάθειας είναι οι ξένες εταιρείες και οι περισσότερες ε, επιδοτήσεις που λαμβάνουμε ουσιαστικά για αυτή τη γη πηγαίνει σε ξένες επιχειρήσεις. Πρέπει λοιπόν να διασφαλίσουμε την παραγωγικότητα της γης και αυτή η παραγωγικότητα να είναι προϋπόθεση για την ε, για να δοθούν επιδοτήσεις. Πρέπει λοιπόν να υπάρχουν συγκεκριμένοι όροι και προποθέσει, αλλά να μην αποκλείονται, να μην εξαιρούνται ε, αυτές οι εκτάσεις από τις επιδοτήσεις. Ευχαριστώ κύριε Σφελάντα. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Και βεβαίω συμμερίζομαι τα συμπεράσματα του εισηγητή για την ε, ανάπτυξη δραστηριότητα ε, και εγκαθίδρυση νέων ε, γεωργών. Είναι πολύ υψηλό το κόστος της γης, όντως. Αλλά για μένα δεν αρκεί, δεν εξαντλείται εκεί η διαπίστωση, γιατί έχουμε να κάνουμε ένα πραγματικό πρόβλημα σχετικό με τη γεωργική κρίση, που είναι η περιορισμένη αποδοτικότητα των εκμεταλλεύσεων. Δηλαδή, αν δεν μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτό το στάδιο τη διάγνωση ενό προβλήματο ω μόνο προβλήματο τη εγκατάσταση νέων γεωργών, δεν θα έχουμε λύσει το πρόβλημα, γιατί ο νέο γεωργό, ο οποίο αναλαμβάνει ένα δάνειο σχέση με την τραπεζά του, χρειάζεται και εγγύησει. Και το βλέπουμε αυτό οι νέοι άνω των 50% δεν είναι διατεθειμένοι να αναπτύξουν γεωργική δραστηριότητα. Και αυτό κρύβει πίσω του ένα μεγάλο οικονομικό πρόβλημα, ότι δεν υπάρχουν διέξοδοι οικονομικές ε, για την γεωργία. Χρειάζεται δηλαδή ένα ολόκληρο πλέγμα δραστηριοτήτων και μετατροπής, ε, επεξεργασίας κτλ. των προϊόντων, ώστε να στηριχθεί η δραστηριότητα γεωργική στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ο κύριος Δέσσε έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ τον ε, εισηγητή για την πρότασή του. κύριο Ρονομέλο με παρακάλεσε να ε, τοποθετηθώ, να, εκφράσω δηλαδή τις δικές του θέσεις. Είναι σκιώδης ο δεν μπόρεσε να είναι παρόν. Μου έχει δώσει το έγγραφό του ε, δεν θα σας το διαβάσω όμως γιατί θα χάναμε τουλάχιστον τρία λεπτά για να το διαβάσω. Πάντως ε, λέει εν ολίγη ότι ως και ο πρόκειται να καταθέσει εκ μέρου τη ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο ορισμένες τροπολογίες ε, για να υπογραμμίσει τη σημασία του μέλλοντο του γεωργικού τομέα ε, και τις ε, αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε αυτό θα σημειώσω ιδιαιτέρως διότι υπάρχουν πολύ διαφορετικές καταστάσεις σε επίπεδο κρατών μελών. Εμείς, η παραδείγματι στη Γερμανία, έχουμε αρκετούς νέους γεωργούς Η ιδέα διαδικασία Omnibus που ανέφερε η κυρία Χεράντς επιτρέπει ένα σχετικά ευρύ περιθώριο ε, δραστηριότητας για τα κράτη-μέλη. Αφήνει αρκετή διακριτική ε, ευχαίρεση στα κράτη-μέλη που θα πρέπει να αξιοποιηθεί πλέον. Έχουμε δυνατότητες λοιπόν και πρέπει να τις αξιοποιήσουμε. Στον κοινωνικό τομέα. Πιστεύω ότι θα πρέπει να του δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση. Εμείς ε, στη Γερμανία, αλλά και σε άλλα κράτη ενδεχομένως, βλέπουμε ότι πιο ηλικιωμένοι γεωργοί μπορούν να μείνουν ε, μέχρι μια πιο προχωρημένη ηλικία ε, για τη συνταξιοδότηση. Φερρυπίν αντί να φύγουν στα 65 από τη γεωργική δραστηριότητα και να παραδώσουν έτσι τη γεωργική του εκμετάλλευση, φεύγουν στα 70 γιατί δεν μπορούν νωρίτερα να εισπράξουν τη σύνταξή του Επειδή είναι οργανωμένο έτσι το συνταξιοδοτικό σύστημα, δεν μπορούν να εισπράξουν σύνταξη νωρίτερα. Αυτό λοιπόν ίσως να απο... αν το αναλάζαμε τα σχετικά συστήματα, ίσω να αποδέσμευε την ε, γεωργική γη και ταυτόχρονα πρέπει να κοιτάξουμε ποια είναι τα νομικά πρόσωπα που έχουν ε, την διακράτηση της γης, κεφαλαιουχικές σε παραδείγματι ε, επιχειρήσεις και όχι ενώσεις προσώπων. Ε, αυτό λοιπόν για τη Γερμανία. Για τη Γερμανία όπου θα πρέπει να αλλάξουν κάποια πράγματα στην νομοθεσία ώστε να αποδεσμευθεί η γεωργική γη από τις μεγάλες επιχειρήσεις και να καταστεί προσβάσιμη και για τον νέο γεωργό. Ευχαριστώ κύριο Σάνι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον ε, Νικόλα Καπούτο, όπως και οι συνάδελφοι. Είναι πραγματικά εξαιρετική έκθεσή του και προσπαθεί να συνοψίσει όλες τις ιδέες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπέρ των νέων αγροτών. Επίσης ε, προτείνει και κάποιες νέες πρωτοβουλίες και σε αυτές θα ήθελα να σταθώ και εγώ. Εδώ και δεκαετίες η κοινή γεωργική πολιτική συνεχιζόταν με ένα ιδιάζοντα τρόπο. Πιστέψαμε ότι αν δώσουμε χρήματα των φορολογουμένων στη γεωργία θα ανθίσει αυτή. Δεν ισχύει όμως αυτό. Χρειαζόμαστε νέα προσέγγιση, νέες πρωτοβουλίες και γι' αυτό συμφωνώ με τον κύριο Μπόγκοβιτς και την επιχειρηματολογία του θα πρέπει να θετήσουμε μια πιο έξυπνη προσέγγιση, ευφυή προσέγγιση. Και έξυπνη προσέγγιση εδώ σημαίνει πώς θα κάνουμε τη ζωή στην Ήπεθρο ελκυστική για τους νέους. Γιατί τα οικονομικά κίνητρα, οι χρηματοδοτικές πρωτοβουλίες από μόνες τους, τα χρήμα από μόνο του δεν μπορεί να λύσει το ηλικιακό πρόβλημα, το ζήτημα της ανανέωσης των γενεών. Θα πρέπει να ε, ενισχύσουμε τις υποδομές, σχολεία, νοσοκομεία, να έχουμε πολλές πρωτοβουλίες ε, στις τοπικές κοινότητες. Μόνο έτσι θα σκεφτούν οι νέοι. Α, γιατί να μην διαλέξουμε τη ζωή στην Ήπεθρο και την ενασχόληση με τη Γεωργία. Επίσης, μιλούμε συνεχώς για τη Γεωργία. Όταν όμως ε, θέλουμε μια έξυπνη προσέγγιση, θα πρέπει να είναι μια νέα προσέγγιση που θα εδράζεται μεν στη Γεωργία, αλλά όχι αποκλειστικά στη Γεωργία. Ευχαριστώ. Και τώρα θα δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον ε, κύριο Χανιώτη. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Oh, thank you. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομος. Πρώτον, θα ήθελα και πάλι να επισημάνω πόσο σημαντική προτεραιότητα είναι από την πρώτη μέρα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η γενολική ανανέωση του ιδιωτικού τομέα. Δεύτερον, οι περισσότερες από τις ε, προτάσεις ε, της έκθεσης ε, πραγματικά είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτε και συνάδουν και με το δικό μας σκεπτικό. Τρίτον, θα ήθελα να σταθώ όχι μόνο στο θέμα της γη, αλλά και στα άλλα ζητήματα που θίξατε. Συνταξιδοτικά συστήματα, φορολόγηση, ιδικτουσιακό καθεστώς κληρονομικό δίκαιο. Μία από τι αλλαγέ που θα επιφέρουμε με τη νέα κοινή γεωργική πολιτική είναι αυτή η διασύνδεση μεταξύ των ε, μέτρων που υιοθετούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ε, εθνική νομοθεσία που διαφέρει σε πολλού ε, τομεί που επηρεάζουν του νέου γεωργού. Αυτό είναι το μοναδικό που θα ήθελα να επισημάνω, ότι είναι ένα από τα βασικά στοιχεία που θα θέλαμε ε, να επιλύσουμε καθώς θα προετοιμάσουμε την αξιολόγηση δικτύπου για τη μελλοντική κοινή γεωργική πολιτική και σίγουρα θα έχουμε και άλλες ευκαιρίες στο μέλλον. Μέχρι τότε σας ευχαριστώ για τις προτάσεις σας. Σας ευχαριστούμε κύριε Θυντά. Και τώρα θα ξαναδώσουμε το λόγο στον εισηγητή μας, τον κύριο Καπούτο, αλλά παρακαλώ χρόνου φίδου. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Άξιον πολύ μεγάλη προσοχή τη παρεμβάση των συναδέλφων και χαίρομαι ιδιαίτερω διότι θα μοιραστώ μαζί τους αυτή την πορεία που θα μας οδηγήσει σε ένα θετικό οπωσδήποτε αποτέλεσμα για τον τομέα μας. Αποδέχομαι και κάποιες οπωσδήποτε πιο επικριτικές ε, διαπιστώσεις, ε, τοποθετήσεις. Είμαι βέβαιος πάντως ότι θα μπορέσουμε στις επόμενες εβδομάδες να βρούμε την χρυσή τομή, μια σωστή λύση έτσι ώστε να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ένα πιο ευνοϊκό περιβάλλον για τους νέους μας, ε, για τη γεωργία. Θα ήθελα πάντως να μιλήσω ιδιαίτερα για την σημασία του ρόλου του νομοθέτη και της Επιτροπής μας, γιατί όταν μιλούμε για νέους πρέπει να είμαστε πιο φιλόδοξοι πιστεύω και να ε, πετάξουμε πιο μακριά την μπάλα στο μέλλον για να ευνοήσουμε ακριβώς και να εξασφαλίσουμε το μέλλον για τον τομέα μας ο κύριος Βίτερμαν σε παραδείγματι για μια φορολογία στοχευμένη σε ε, αποτελέσματα αλλά και τον Σάνι και άλλων για την ευφυή προσέγγιση όπως θα την ονόμασα μια ευφυή προσέγγιση για τη γεωργία είναι στοιχεία ε, θεμελιώδη που θα πρέπει οπωσδήποτε να χαρακτηρίζουν όλη μας τη δραστηριότητα και τις επιλογές. Βεβαίως όλες οι άλλες προτάσεις είναι πολύ σημαντικές. Ε, θα τις συμπεριλάβουμε στις εντατικές εργασίες που θα ακολουθήσουν τις επόμενες ημέρες, στις οποίες και θα αφιερώσω εγώ προσωπικώς μεγάλο μέρος των δραστηριοτήτων μου προκειμένου να εξασφαλίσω μια συνθετική πρόταση, μια πρόταση που να είναι ικανοποιητική για όλους τους συναδέλφους. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Μας είπατε για, τις, ε, για την προθεσμία για τις τροπολογίες που λήγει στις 19 Ιανουαρίου. Οπότε ολοκληρώνουμε το σημείο 4 και περνάμε στο σημείο 5 της ημερήσιας διάταξης. Όπως ε, ξέρετε, στις 10 με 13 Δεκεμβρίου έλαβε χώρα στον Πένος Άιρες η 11η Υπουργική Διάσκεψη ε, της Παγκόσμιας Οργάνωσης Εμπορίου και κατέτηση των συντονιστών της Επιτροπής Γεωργίας ε, αποφασίσαμε να συμμετέχει και ένας εκπρόσωπος της Επιτροπής μας στην αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να μην έχουμε μόνο εκπρόσωπο της Επιτροπής Εμπορίου. Ο εκ μέρους μας λοιπόν πήγε η κυρία Μαγκίνες, αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ως τέτοια ήταν και επικεφαλής ε, της αντιπροσωπείας μας, ε, εκπροσωπώντας ιδιαίτερα τη Γεωργία. Ε, αδυνατή να είναι στην αίθουσα η κυρία Μαγκίνες αυτή τη στιγμή, αλλά τη βλέπουμε, χάρη στην τεχνολογία θα έχουμε μία σύνδεση με βίντεο διάσκεψη, τηλεδιάσκεψη μαζί της για να μας παρουσιάσει τα αποτελέσματα της εκτιμής της και την διεξαγωγή αυτής της ε, υπουργικής διάσκεψης και των άλλων συναντήσεων στις οποίες έλαβε μέρος. έγιναν πολλές διμερείς επαφές για θέματα εμπορίου. Μάλιστα έχετε λάβει και τη γραπτή έκθεση της ε, κυρίας Μαγκίνες από τον Buenos Άιρες. Θα ακούσουμε όμως ε, την ίδια την κυρία Μαγκίνες που θα μας ενημερώσει. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Καλημέρα σας κύριε Πρόεδρε, καλημέρα αγαπητοί συνάδελφοι και σας ευχαριστώ που κατεξαίρεση επιτρέψετε τηλεδιάσκεψη ε, γιατί χρειάστηκε να μεταβώ κατεπηγόντως στο Δουβλίνο για μια κηδεία. Θα σας παρουσιάσω τα αποτελέσματα των συζητήσεων ε, του Buenos Aires. Καταρχήν ήταν πολύ καλή ιδέα των συντονιστών της Επιτροπής Γεωργίας να έχουμε και ένα δικό μας εκπρόσωπο και για τις άτυπες επαφές, αλλά και για το επίσημο σκέλος των συζητήσεων ε, της Παγκόσμιας Οργάνωσης Εμπορίου. Καταρχήν έγινε και μια κοινοβουλευτική διάσκεψη του ΠΟΕ και συμμετείχα εκεί ως αντιπρόεδρος στην έναρξη και στη λήξη. Μιλήσαμε για τα, την ισότητα των φύλων, το εμπόριο γενικά, αλλά η βασική μας ανάγκη ε, ήταν να λάβουμε μέρος στην υπουργική διάσκεψη και ήταν μεγάλες οι προσδοκίες από την έκβαση αυτής της υπουργικής διάσκεψης. Αν θυμάστε όμως τα σχόλια μετά την ολοκλήρωση της διάσκεψης από τους Επιτρόπους Χόγκαν και Μάστρομ θα διαπιστώσετε ότι εξέφρασαν την απογοήτευσή τους για την ελάχιστη πρόοδο που σημειώθηκε. Εμείς φανταζόμασταν και είχαμε πολύ ψηλότερες προσδοκίες. Ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε είναι πώς θα προχωρήσουμε από εδώ και πέρα. Ε, εν είδη να σα πω ότι η κοινή γεωργική πολιτική στο πλαίσιο του ΠΟΕ και συμφωνώ με τη συζήτηση που κάνατε και την ενδιαφέρουσα έκθεση του Καπούτα για τους ε, νέους αγρότε, Η κατάσταση στη γεωργία άλλαξε ε, λόγω του ΠΟΕ και της ανάγκης να καταργηθούν οι στρεβλωτικές του εμπορίου επιδοτήσεις και μάλιστα ο πρόεδρος ε, της ε, Επιτροπής Γεωργίας του ΠΟΕ με ενημέρωσε για την εντύπωση που έχουν παγκοσμίω για την Ευρωπαϊκή Γεωργία. Βέβαια αναγνωρίζουν ότι η Ευρώπη άλλαξε τη γεωργική της πολιτική ώστε να μην στρεβλώνει τόσο πολύ το εμπόριο γιατί έχουμε αποσυνδέσει πλέον τις ενισχύσεις αλλά από τις ε, συζητήσεις που έγιναν για τους νέους αγρότες προέκυψαν άλλα ζητήματα που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Πάντως κάποια κράτη-μέλη της, του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου θεωρούν ότι εξακολουθούν να είναι απαράδεκτα και υπερβολικά τα επίπεδα επιδοτήσεων που εφαρμόζουμε στην κοινή γεωργική πολιτική στο μπλε και πράσινο κουτί. Αναγνωρίζουν την πρόοδο μα, αλλά θεωρούν ότι θα πρέπει να σημειώσουμε ακόμη μεγαλύτερη πρόοδο στον περιορισμό των επιχορηγήσεων. Ένα άλλο θέμα που συζητήσαμε ήταν η παράνομη αλληλεία και οι επιδοτήσει ε, στο βαμβάκι και άλλε επιδοτήσει κατά την έναρξη της υπουργικής διάσκεψης που ήταν πολύ εντυπωσιακή, πολύ επίσημη και πανηγυρική, ήταν πολύ καλή διοργάνωση και κατά την έναρξη λοιπόν η Βραζιλία, Αργεντινή, Ουρουάη και Παραγουάη παρουσίασαν την διακήρυξη του Buenos Aires με στενή δεσμευση υπέρ του ελευθέρου εμπορίου και της πολυμέρειας καλώντα και τα υπόλοιπα κράτη να προσχωρήσουν. Και αυτή ήταν μια προσπάθεια για να προσελκύσουν την υποστήριξη και των Πολιτειών και ένα άλλο χώρο. Κάτι που δεν συνέβη, γιατί η παρέμβαση των Πολιτειών, όπως αναμενόταν υποστήριξε μεν τον ΠΟΕ, αλλά εξέφρασε σοβαρές ανησυχίες για την κατεύθυνση που παίρνει. Επίσης, ε, επισημάνθηκε η ανάγκη να σημειωθεί πρόοδος, αλλά τελικά δεν στέφθηκε με επιτυχή η εμπορική διάσκεψη, δεν σημειώθηκε ε, σημαντική πρόοδος ε, στα ζητήματα που συζητήθηκαν και αυτό το σήμανε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και επίσης υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι άτυπο μέσα στην ε, πρόταση που παρουσιάστηκε από τον συνάδελφο που ήταν μαζί μου το υπέβαλε. Ήταν πολύ σημαντικές και οι άτυπες συναντήσεις πρέπει να πω. Ιδιαίτερα ε, τα θέματα που έχουν να κάνουν με τη Συμφωνία Εμπορίου με Μερκοσούρ και την αντιπαράθεση. Ε, στο Βουένος Αέρες είχαμε την ευκαιρία να διαπιστώσουμε δυνατότητες για εξελίξεις. Δεν τις ε, είδαμε ακόμη να υλοποιούνται, αλλά διαπιστώνουμε και θεωρούμε ευπρόσδεκτο το γεγονός ότι η Αργεντινή, η Παραγουάια, η Βραζιλία προσπαθούν να πιέσουν ώστε να υπάρξει μια κάποια πρόοδος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως θέλει συμφωνία με τη Μερκοσούρ και αυτό βέβαια ιδιαίτερα για το Βόιο έχει τη σημασία του για την ε, Επιτροπή Γεωργίας, η Κορζικά, ε, Γάλλοι, ε, παραγωγή Βόιου κρέατος αλλά και Ιρλανδοί ήταν παρόντες στο Buenos Aires και υπεγράμμισαν τη σημασία μιας καλής συμφωνίας. Εν όλο λοιπόν οι ευκαιρίες που δόθηκαν για συνομιλίες στο Buenos Aires για το εμπόριο σε γεωργικά προϊόντα ήταν πολύ καλές και χρήσιμες για τον ε, ΠΟΕ και τις περαιτέρω εξελίξεις. Εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση θα, πρέπει να προσπαθήσουμε να τον ενισχύσουμε, πιστεύω, γιατί κάποιοι προσπαθούν να τον αποδυναμώσουν και οπωσδήποτε σε θέματα που έχουν να κάνουν με την Ινδία, από θέματα σε τρόφιμα, ασφάλεια επιστηστική, δεν είδαμε να υλοποιείται η πρόοδος που περιμέναμε, που επιδιώκαμε λόγω της τάσης των ΗΠΑ. Ο ΠΟΕ λοιπόν ως θεσμός αλλά και ως δομές πρέπει να ενισχυθούν και είναι προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης να το πράξουμε αυτό. Πρέπει επίσης ε, να παρακολουθήσουμε μαζί με τους συναδέλφους τις εξελίξεις στη Μερκοσούρ και θέλω να ευχαριστήσω βεβαίως ολοκληρώνοντας όλους αυτούς και από την Επιτροπή Εμπορίου αλλά και από την Επιτροπή Γεωργίας τους συναδέλφους και το προσωπικό που υποστήριξαν και διευκόλυναν την οργάνωση. Τελευταίο σήμερα, σήμερα θα ε, είμαι στην κηδεία του Πίτερ Σάδελαντ πρώην ε, Επιτρόπου Γεωργίας αλλά ταυτόχρονα και Γενικού Γραμματέα στην ΚΑΤ και τον ΠΟΕ. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα σημάδι για το τι μπορούμε να κάνουμε και το τι πρέπει να κάνουμε, να εργαστούμε δηλαδή επικοδομητικά ως Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε ο ΠΟΕ να λειτουργεί αποτελεσματικά και να μην επιτρέψουμε να αποδυναμωθεί στο μέλλον. Αυτά, Πρόεδρε, και περιμένω τις ερωτήσεις των συναδέλφων. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε σύντομοι και αποτελεσματικοί. Και μάλιστα το ζήτημα αυτό εξετάζεται και στην Επιτροπή Εμπορίου και ήταν σημαντικό να ακούσουμε και τη γνώμη της ε, Επιτροπής Εμπορίου και καλό να συνεργαστούμε με την Επιτροπή Εμπορίου, ώστε να προσφέρουμε και τη δική μας τη γεωργική διάσταση. Γιατί ε, δεν έχουν ε, μεγάλη γνώση για την Επιτροπή Γεωργίας η Συνάρτηση Επιτροπής Εμπορίου. Θα πρέπει εμείς να προσθέσουμε αυτή τη γεωργική διάσταση. συναρτηση της Επιτροπής Εμπορίου. Θα πρέπει εμείς να προσθέσουμε αυτή την γεωργική διάσταση. Η κυρία Σκοτ Κάτω. Γεια σου Μαρέτ και ευχαριστώ πολύ για την ξεκάθαρη αυτή παρουσίαση. Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων ε, στη Μερκοσούρ υπήρξαν κάποιες συνδέσεις με την Greenpeace και για τις κάτω χώρες που ενέχουν ε, στοιχεία προβληματισμού ε, για τους γεωργούς μας, ιδίως εάν υπάρχουν χαμηλά πρότυπα περιβαλλοντικά από την άλλη πλευρά. Αυτό είναι του ανταγωνισμός για τους δικούς μας γεωργούς. Ε, σε ό,τι αφορά την επίλυση διαφορών ε, μεταξύ κρατών, αυτό σημαίνει ότι δεν θα είναι μη, ε, κάτι που θα μπορεί να επιβληθεί. Ε, Ιδίω ό,τι αφορά την υποψήφιση των δανειστών στη Βραζιλία, υπάρχει έλλειψη και τη αρχή τη προφύλαξη για του απαρκεί ε, ελέγχου για την υγεία των ζώων και ε, ε, ανεπαρκής ε, έλεγχους για τα ζανιοκτώνα. Ποιε είναι οι δικές σου σκέψεις σε ό,τι αφορά τις συζητήσεις κατά τις διαπραγματεύσεις και κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εκδώσει, θα δημοσιοποιήσει την εξολόγηση αντικτύπου για τις πιθανές προϋποθέσεις βιωσιμότητας. Ε, επίσης με ενδιαφέρει ε, τι, συνέβη και δεν επετράπη η είσοδο στην Αργεντινή σε πολλέ Η Επίτροπο Μάλστρομ βέβαια αντέδρασε έντονα, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο υπήρξαν κάποιε άλλε επιπτώσει. Και τέλο, <clears throat> υπήρξε έλλειψη τελική διακήρυξη ε, του ΠΟΕ. Αυτό δείχνει ότι τα, το πολιτικό σχέδιο ήταν αρκετά δύσκολο. Ιδίω στο πλαίσιο του Brexit μα ενδιαφέρει αυτό. Σαφώ και ε, όσοι είναι υπέρ του Brexit λένε δεν υπάρχει πρόβλημα, θα ακολουθήσουμε του κανόνε ΠΟΕ. Όμω αυτό από πολιτική άποψη θα είναι πολύ πιο δύσκολο από ό,τι περίμεναν. Πρέπει να φύγω τρέχοντα προ την ε, Επιτροπή ΕΚΟΝ. Ευχαριστώ λοιπόν εκ των προτέρων, ακόμα και αν δεν θα είμαι εδώ στι απαντήσει. Ευχαριστώ. Παρακαλώ να περιστείτε στην υποβολή ερωτήσεων. Για... Βέβαια μπορεί να χρειάζονται και τα σχόλια από και που, αλλά 1,5 λεπτό έχει ο καθένα καλύτερα να περιοριστεί στις ερωτήσεις. Μέρετ, θέλω και εγώ να εκφράσω θερμές ευχαριστίες για την συμμετοχή στην διάσκεψη αυτή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να είναι παρούσα η Επιτροπή Γεωργίας ε, στον ΠΟΕ. Πρόκειται για διαπραγματεύσεις που έχουν πολύ μεγάλη σημασία για μας. Η Ευρωπαϊκή Γεωργία να κερδίσει εάν μπορούμε να προχωρήσουμε ενωμένοι και δεν κάνουμε χωριστές συμφωνίες με τη Μερκοσούρα αλλά μόνο μέσα από το πλαίσιο του ΠΟΕ μεριμνούμε για συμφωνίες οι οποίες ασφαλώς ε, έτσι θα λαμβάνουν υπόψη και τη δύναμή μας ε, μεγέθη και δεν επιτρέπουν την ε, στρέβλωση του εμπορίου. Έτσι λοιπόν θα είναι σημαντικό να έχουμε μια έκθεση πρωτοβουλίας ε, όχι μόνο για την Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Μπερκοσούρα αλλά ταυτόχρονα και ε, μια δουλειά κοινή με την Επιτροπή Εμπορίου που θα ε, δίνει τις πιο πρόσφατες εξελίξεις. Δεν πρέπει η Ευρώπη εδώ να παρασυρθεί σε διμερείς χωριστές συμφωνίες. Είναι σημαντικό για μένα να προχωρήσουμε στις διαπραγματεύσεις του ΠΟΕ να συμμετάσχουμε και κύριε Πρόεδρε δεν ξέρω εάν υπάρχει η δυνατότητα για μια κοινή συζήτηση με την Επιτροπή Εμπορίου για αυτές τις διαπραγματεύσεις ε, του Μπόνα Aires ώστε να ε, διατυπώσουμε με, σαφής, ε, με σαφή τρόπο και τις θέσεις της Επιτροπής Γεωργίας. Ευχαριστώ κύριε Σοραπέ. Και θα ήθελα στη γραμματεία να ζητήσω να αναλάβει τις σχετικές ε, εργασίες. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χαίρομαι ιδιαίτερω που η Επιτροπή μα ε, εκπροσωπήθηκε σε αυτέ τι συζητήσει. Είναι πολύ συγκεκριμένο αυτό ο τομέα τη γεωργία, γιατί λαμβάνει επιδοτήσει και διαφορετικέ μορφέ επιδοτήσεων ε, ανάλογα με την ε, περιοχή του κόσμου. Οι διεθνεί συμφωνίε είναι πολύ σημαντικέ. Από την άλλη όμω, αν δούμε την ΣΥΤΑ, μιλήσαμε για το κατά πόσο είναι δίκαιη Πρέπει λοιπόν αυτές οι συμφωνίες να είναι ωφελείς για όλους. Όμως ε, σήμερα δεν είμαστε σίγουροι ότι ισχύει αυτό και δεν είμαστε σίγουροι ότι θα είναι επωφελής ε, αυτές τις συμφωνίες που έχουμε υπογράψει προς τους γεωργούς. Ε, ενδεχομένως μόνο ο εμπορικός τομέας να επωφεληθεί και όχι ο γεωργικός. Γιατί θα ανέβουν και οι εμπορικές τιμές. Άλλη πτυχή τώρα, η ανταγωνιστικότητα κατά την εισαγωγή εμπορευμάτων. Είναι πολύ σημαντικό να διασφαλίζουμε ότι τα προϊόντα αυτά έχουν παραχθεί με βάση τις ίδιες ε, τεχνολογικές και περιβαλλοντικές και άλλες ε, διατάξεις που ισχύουν για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ιδάλλως θα είναι αθέμητος ανταγωνισμός και δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε. Βλέπουμε ότι κάποιες χώρες θέλουν ε, να εξαγάγουν ενέργεια χωρίς να πληρούν τις περιβαλλοντικές προδιαγραφές και έτσι και εμεί θα πρέπει να επιμείνουμε ιδιαίτερου στις περιβαλλοντικές διαστάσεις. Ο κ. Φλάνναγκαν, ευχαριστώ. Καλή χρονιά Μερίτ και καλή ε, επιτυχία με τις προσπάθειές του σε ό,τι αφορά την Ελλαδική Προεδρία βάσει ιστορικών δεδομένων και των περιβαλλοντικών ε, τις πληρωμές Green Box. Υποτίθεται ότι είναι πληρωμές και επιδοτήσεις που δεν ε, στρεβλώνουν την αγορά και αφορούν τα έτη αναφοράς 2000-2002. Έχουν λάβει την έγκριση του ΠΟΕ. Ποια είναι η γνώμη σου. Ευχαριστώ κύριο Σάγνιου. καλημέρα, καλή χρονιά και σας ευχαριστούμε για την πολύ καλή αυτή παρουσίαση και σε λυπητήρια. Πολύ απλό το ερώτημα. Έθεσε κανείς το ερώτημα της δημικροβιακής αντοχής ε, στους, ε, στις συζητήσεις αυτές υπό τον ΠΟΕ. ΠΟΕ. Ε, υπάρχουν χώρες που θέλουν να παρεμποδίσουν τους γεωργούς σε ό,τι αφορά την χρήση τέτοιων αντιβιωτικών. Από την άλλη όμως δεν έχουν πρόβλημα να εισαγάγουν προϊόντα τέτοια. Ευχαριστούμε πολύ να δώσουμε το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα από την DG Agri. Παρακαλώ. Thank you, sir. I can be... Ευχαριστώ πολύ σύντομα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σαφώς ε, και απογοητεύεται ε, και εκφράζει την απογοήτευσή τη ε, λόγω τη έλλειψη διακήρυξη στο τέλο. Δεν προκαλεί έκπληξη, γιατί εκ των προτέρων έχουμε καταλάβει ότι θα είναι πολύ δύσκολη διαδικασία και η Επιτροπή και η, εκπροσ... η Αντιπροσωπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν πολύ καλά προετοιμασμένη. Έχει συμμετάσχει ενεργά στις ε, ε προπαρασκευαστικές εργασίες. Νομίζω ότι ήταν θετικός ο ρόλος Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και αυτό αναγνωρίζεται ευρέως. Ε, εμείς τουλάχιστον δεν ξεπεράσαμε, δεν έχουμε υπερβεί τις κόκκινες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορούμε από την άλλη να πούμε ότι υπήρξε πολύ καλή συνεργασία μεταξύ Επιτροπής, ε, Κοινοβουλίου και κάτων μελών. Από εδώ και πέρα πρέπει να μας προβληματίσει αυτό το ζήτημα, να δούμε τυχόν ε, μελλοντικά βήματα και κινήσεις, να δούμε ε, πώς μπορούν να επανεκκινήσουν οι διαπραγματεύσεις ε, στο γειτονικό τομέα, να εξετάσουμε και νέες ε, προσεγγίσεις και να βασιστούμε και στα επιτεύγματα του παρελθόντος, όπως η απόφαση που είχε υιοθετηθεί στο Ναϊρόμπι. Τα πράγματα ενδεχομένως να επιδεινωθούν πριν βελτιωθούν Οπότε εμείς ε, θέλουμε να συνεχίσουμε την επικοδομητική μας προσπάθεια στις ε, διαπραγματεύσεις υπό τον ε, ΠΟΕ για να περασπιστούμε όσο μπορούμε καλύτερα τα ευρωπαϊκά συμφέροντα και αν αυτό καταστεί δυνατόν να ενισχύσουμε το πολυμερές σύστημα διαπραγματεύσεων. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Μπορείτε να τις αποστείλετε και μέσω mail προς τη γραμματεία. Τώρα θα ήθελα να δώσουμε το λόγο και πάλι στην κυρία Μαγκίνες για να απαντήσει. Thank you, Chair. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ για τα σχόλια και τις ερωτήσεις. Όντως είχαμε μια πολύ καλή ενημέρωση, ένα έγγραφο πολύ καλό ενημερωτικό από τον Φιλίπ Μουστάχ, πολύ σημαντικό αυτό να το λάβουν υπόψη οι συνάδελφοι. Επίσης θέλω να σημειώσω ότι απαρτίζεται από 164 χώρες ΠΟΕΤ, ότι δεν είναι ευχερής η διαδικασία, δεν νομίζω ότι τα ξαφνιάζει κανέναν. Ωστόσο ε, το, το πρόβλημα είναι ότι οι μεγαλύτεροι παράγοντες αυτής της διαδικασίας δεν συνεργάζονται όπως θα θέλαμε. Εκεί ακριβώς εντοπίζεται το πρόβλημα και πρέπει να μεριμνήσουμε ώστε να λάβουμε δράση για τα πράγματα ενδέχεται να χειροτερέψουν πριν ε, βελτιωθούν, αν και πάντα η ελπίδα είναι ότι θα βελτιωθούν. Για το Μερκοσούρ δεν, είχε, δεν ήταν στο επίκεντρο των συζητήσεων, στο περιθώριο μόνο μπόρεσε η Ευρωπαϊκή Αντιπροσωπεία να αναπτύξει συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κάποιες οργανώσεις με κυβερνητικές και άλλες από τη Μερκοσούρ. Σημασία βέβαια έχουν οι προδιαγραφές, τα πρότυπα και η ανάγκη για προστασία και τήρηση των ευρωπαϊκών πρωτήτων, αλλά και ζητήματα του ανταγωνισμού. Για το δεύτερο ερώτημα, για τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις και τον αποκλεισμό τους, ε, ήταν ε, εμφανείς οι διαμαρτυρίες γύρω από τους χώρους του ε, της διάσκεψης ε, ειρηνικές διαμαρτυρίες και αυτό επίσης αξιολογήθηκε θετικά αλλά και βεβαίως η κυρία Μάλστρομ η Επίτροπος υπεγράμμισε την ανησυχία της για την δυνατότητα να συμμετέχουν οι κυβερνικές οργανώσεις που έχουν τόσο σημαντικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία. Ε, από εδώ και μπρος ΠΟΕ και πάντα ε, έχοντας υπόψη τον Brexit ε, έχουμε να πούμε τα εξή. Παρουσία του Βασιλείου, η παρουσία του Ηνωμένου Βασιλείου ήταν ορατή και οι συναδέλφοι από το Ηνωμένο Βασίλειο πάντα ε, τοποθετήθηκαν με ε, το μάτι στραμμένο στις προοπτικές του Brexit και τις εξελίξεις αυτές. Ε, πάντως, το Ηνωμένο Βασίλειο υπέδειξε πως ε, θα παραμείνει πιστό στις αρχές του ΠΟΕ και ότι δεν θα υπάρξουν προβλήματα ως προς αυτό ταυτόχρονα ποσοστώσεις και άλλα ζητήματα πρόσβασης που είναι πολύ περίπλοκα δεν έχουν κλείσει γιατί ο ΠΟΕ δεν έχει δώσει ακόμη το πράσινο φως για τα όσα επιδιώκουν Ηνωμένο Βασίλειο και Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κυρία Μίλλερ επίσης διατύπωσε παρατηρήσεις για τον ΠΟΕ. Δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω με τις δικές της παρατηρήσεις. Αν δεν υπήρχε ο ΠΟΕ δηλαδή θα καταλήγαμε σε πολέμους εμπορικούς. Ένας από τους συναδέλφους από την Επιτροπή Εμπορίου, ο κύριος Ρούμπιχ άλλωστε, το στις τοποθετήσεις του ε, μετά από την Υπουργική Διάσκεψη ε, και είπε εμπορικός πόλεμος ίσον πόλεμος, ένοπλη σύραξη. Γι' αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό να τους αποφύγουμε. Είναι επίπονη η προσπάθεια να διατηρηθεί ο διάλογος σε επίπεδο ΠΟΕ για να αποφύγουμε περαιτέρω και πολύ σκληρές αντιπαραθέσεις. Για τον κύριο Φλάναγκαν και τις σκληρές παρατηρήσεις του θέλω να ασχολιάσω μόνο το εξή στην ερώτηση του τι πιστεύω εγώ. Οι ιστορικά, οι συνδεδεμένες ε, πληρωμές ενισχύσεις ε, υφίσταται για να διατηρηθεί ένα σύστημα το οποίο προϋπήρχε. Δεν μπορούν όμως να συνεχιστούν επαόριστον, το γνωρίζουμε όλοι αυτό. Θα πρέπει να βρούμε ένα νέο σύστημα με βάση τις προτάσεις που υπάρχουν που θα εξασφαλίζει και την παροχή του δημόσιου αγαθού αλλά και τον θεμητό και ισότιμο ανταγωνισμό. Για το πράσινο κουτί δεν μπορώ να απαντήσω εγώ. Είναι αποφάσεις του ΠΟΕ οι οποίες λαμβάνονται και σε σχέση με τις αποσυνδεδεμένες ε, πληρωμές. Μέχρι εκεί θα φτάσουν τα σχόλιά μου για τον κύριο Άγνιου εν για την αντιμικροβιακή αντίσταση. Είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν γέρθει. Είναι όμως σημαντικό ζήτημα και πρέπει στο μέλλον πιστεύω να τεθεί. Και μια-δύο προτάσεις ακόμη, Πρόεδρε, για να ολοκληρώσω. Όταν οι συναδέλφοι μιλούν ε, για την ε, ανάγκη να συνεργαστούμε και να συνδυάσουμε τι εργασίε μα με αυτέ τη Επιτροπή εμπορίου. Συμφωνώ απολύτω, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Διαπιστώνω ότι στην έλφη από την Επιτροπή Εμπορίου είναι διαθέσιμη σε τέτοια συνεργασία και άλλωστε το δήλωσαν και κατά τι επαφέ που είχαμε στο Buenos Aires. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να επιδιώξουμε συνεργασία μεταξύ διαφόρων επιτροπών για να προωθούμε τι θέσει μα. Γιατί για τα θέματα των νέων γεωργών, για τα θέματα των προβλημάτων ε, που αντιμετωπίζει κάποιο που θέλει να ξεκινήσει μια γεωργική δραστηριότητα και να εγκατασταθεί σε κάποια χώρα ε, είναι όπως και της ε, διαδοχής της, ε, των ποσοστών των νέων στη γεωργία. Όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία μας ενδιαφέρουν και που θα πρέπει να υποστηρίξουμε σε συνεργασία με τους συναδέλφους από την Επιτροπή Εμπορίου. Είναι απόφαση της Επιτροπής μας βεβαίως να προχωρήσουμε σε αυτή τη συνεργασία. Ήταν χρήσιμη πάντως, είναι χρήσιμη και τώρα και θα είναι και στο μέλλον. Και πρέπει πιστεύω να συνεργαζόμαστε και στο μέλλον με συναδέλφους της Επιτροπής Εμπορίου σε τέτοιου είδους αποστολές. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα λοιπόν αυτό να το λάβουμε υπόψη, αυτή την ανάγκη συνεργασίας με την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου που επισημάνατε και εσείς και οι συνάδελφοι. Επίσης, ε, αυτό θα ήθελα να επιθυμίσω στην ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, για το την επιρροή που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη για τις, στις διαπραγματεύσεις ε, ε, και πώς οι υφιστάμενες εμπορικές συμφωνίες αλλά και οι διαπραγματεύσεις για τις μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες πώς θα επηρεάσουν τη Γεωργία. Αυτό το θέμα της επιρροής ε, στη Γεωργία θα πρέπει να το λαμβάνει υπόψη η διαπραγματεύση Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Περιμένουμε φυσικά την επόμενη νομοθετική πρόταση. Πάντως το γενικό συμπέρασμα είναι ότι θα πρέπει να μεριμνήσουμε για αγαστή συνεργασία με τις Επιτροπές Εμπορίου, ΙΜΚΟ, προστασία του Καταναλωτή, περιβάλλοντος και ασφάλειας των τροφίμων, γιατί ε, και σε αυτές υπάρχουν θέματα που συζητώνται και που ενδιαφέρουν και τη γεωργία. Θα πρέπει λοιπόν να, να έχουμε στενή συνεργασία με τις επιτροπές αυτές. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε, αλλά θα πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση για να ενισχύσουμε τις ε, δραστηριότητές μας και σε άλλους τομείς. ιδιαίτερα τώρα που έχουμε ξεκινήσει τη συζήτηση για τη μεταρρυθμίση ΚΑΠ. Και μάλιστα Σάββατο Κυριακή Δευτέρα είχαμε σημαντική διάσκεψη που οργάνωσε ο Επίτροπος Έτιγκερ για τα προβλήματα χρηματοδότησης στις ε, επόμενες ε, δημοσιονομικές προοπτικές μετά το 2020. Ε, αξιοποιήθηκαν όλες οι αίθουσες, ε, υπήρξε και μετάδοση απευθείας, γύρω στα χίλια άτομα συμμετείχαν και είχαμε σχετικά αισιόδοξε ενδείξεις και ειδήσει σε ό,τι αφορά ιδιαίτερα την πολιτική ε, συνοχής και, την πολιτική, και τη γεωργική πολιτική και για την, τις αγροτικές περιοχές και την Ήπεθρο που λαμβάνουν κάποια κονδύλια και από την πολιτική συνοχή. Ευχαριστούμε θερμά τους συναδέλφους, την Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και χαίρομαι που είχαμε τη δυνατότητα να ενημερωθούμε και απευθεία από την κυρία Μαγκίνε. Πάντως θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό σίγουρα. Σα ευχαριστώ. Ολοκληρώνουμε το σημείο 5 και περνάμε στο σημείο 6, τι ενοποιημένες στατιστικέ για τι γεωργικέ εκμεταλλεύσεις. Έλαβε χώρα ο δεύτερος τρίλογος, ανέκυψαν όμω νέα προβλήματα και έτσι δεν τελεσφόρησε ο δεύτερο τρίλογο. Για να επιταχύνουμε όμω τι διαδικασίε, θα δώσω κατευθείαν το λόγο στην κυρία Νταντσίλα, την εισηγήτριά μα, και να μα ενημερώσει εν συντομία για την εξέλιξη στο θέμα αυτό και σε τι φάση της διαδικασίας βρισκόμαστε. Παρακαλώ κύριε Νταντσίλα, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να, να σας ευχαριστήσω και να ευχηθώ σε όλους σας καλή χρονιά. Όπως είπατε κύριε Πρόεδρε, δεν καταφέραμε να ολοκληρώσουμε στο τέλος του 2017 στην τελευταία ολομέλεια του Στρασβούργου ε, να καταλήξουμε σε συμφωνία για το θέμα αυτό. Ε, το ζήτημα αυτό ήταν μέχρι στιγμής ιδιαίτερα τεχνικό, τώρα έχει γίνει ακόμη πιο δύσκολο εξαιτίας του νέου άρθρου 12α που εισήγαγε το Συμβούλιο και αφορά την προστασία των δεδομένων. Πιστεύω παρόλα αυτά ότι καταφέραμε και σημειώσαμε αρκετή πρόοδο στο ζήτημα των ενοποιημένων στατιστικών, αλλά η αναζήτηση της απαραίτητης θεσμικής οροπίας δεν μας επέτρεψε την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων. Ε, το Συμβούλιο φάνηκε τελείως αδιάλακτο και ανένδοτο στη, στις διαπραγματεύσεις και δεν δέχτηκε καμία παραχώρηση ε, σε ό,τι αφορά τα άρθρα 8 και 9. Θα ήθελα παρόλα αυτά να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί η δική της τάση ήταν ιδιαίτερος επικοδομητική ήταν και διαλλακτική και έδειξε πνεύμα συνεργάσιμο και κατανόηση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί πάνω απ' όλα ευελιξία χρειαζόμαστε, ελαστικότητα. Ε, με την Βουλγαρική Προεδρία θα ε, συζητήσαμε τα άρθρα 8 και 9 και εξηγήσαμε στη Βουλγαρική Προεδρία ότι δεν πρόκειται να επιληφθούμε ε, αν δεν έχουμε μια ρεαλιστική εντολή από το Συμβούλιο προς την Βουλγαρική Προεδρία. Σε ό,τι αφορά τώρα τα ιδιωτικά δεδομένα, άρθρο 12, αυτό το πρόβλημα ξεφεύγει από το πεδίο εφαρμογή των γεωργικών ε, στατιστικών και θα δημιουργήσει ε, προηγούμενα και για άλλα στατιστικά στοιχεία που αφορούν τα κοινωνικά ζητήματα, για παράδειγμα. Πάντως θα ήθελα να συνεργαστώ ε, και με τις άλλες επιτροπές για να έχουμε κοινή θέση και να απευθύνω μια έκκληση προς τα μέλη της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ των Πολιτικών Ελευθεριών. Θεωρώ ότι ο γενικός κανονισμός για την προστασία των δεδομένων και οι διατάξεις του είναι επαρκής ως προς την προστασία που εξασφαλίζουν και δεν θεωρώ ότι είναι απολύτως απαραίτητο το νέο άρθρο που προτείνει το Συμβούλιο, το 12α. Ε, πολύ θα ήθελα να είχαμε ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις στη διάρκεια της Εσθονικής Προεδρίας, κάτι που θα διευκόλυνε την κατάσταση στην ε, Ισπανία, Πορτογαλία και Ελλάδα. Γιατί ε, είχαν ζητήσει τρεις χώρες αυτές παράταση μέχρι το 2019. Ελπίζω να ε, διεκπαιρεώσουμε το ζήτημα το συντομότερο δυνατό, αλλά αυτό δεν πρόκειται να γίνει χωρίς να ληφθεί υπόψη και η γνωμοδότηση Επιτροπής Γεωργίας. Ευχαριστώ τους και οδησηγητές, τη γραμματεία, τους συνεργάτες μας για την ε, ανεκτήμητη συνεισφορά τους. Ελπίζω ε, στο μέλλον να είναι καλύτερα τα πράγματα. Δεν καταφέραμε να έχουμε μία πρόοδο με συμπερίληψη των θέσεών μας στη διάρκεια του 2017. Πάντως ελπίζω ότι στη διάρκεια της Βουλγαρικής Προεδρίας τα πράγματα θα είναι πιο αίσια και θα συνεχιστούν οι μέχρι τώρα εργασίες για να καταλήξουν. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε για τις προσπάθειές σας κυρία Νταντσίλα και ευχαριστούμε και τους συνεργάτες σας. Δεν ξέρω αν υπάρχουν ερωτήσεις ε, προς την ε, εισηγήτρια την κυρία Νταντσίλα. Αν ναι, παρακαλώ, μπορείτε να τις υποβάλλετε. Δεν βλέπω ερωτήσεις. Θεωρώ ότι ήταν επαρκής η ενημέρωση δηλαδή της κυρίας Νταντσίλα. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία και καλή συνέχεια κυρία Νταντσίλα. Αν χρειαστεί και στο μέλλον ενημέρωση, μην διστάσετε να μας το επισημάνετε. Σας ευχαριστώ. Περνάμε τώρα στο σημείο 7. την ανταλλαγή απόψεων με τα μέλη της Επιτροπής ε, των Περιφερειών και καλωσορίζω θερμά τα μέλη της Επιτροπής των Περιφερειών και ιδιαίτερα της ε, Επιτροπής για τους Φυσικούς Πόρους. Θα ξεκινήσουμε τη διαβούλευση με την Επιτροπή Περιφερειών. Ο κύριος Όση Μαρτικάινεν, που είναι ο πρόεδρος ε, της Επιτροπής Φυσικών ε, Πόρων, είναι ο πρώτος καλεσμένος μας, καθώς ε, και ο εισηγητής ο κύριος Γκυγιόμ Κρός, αλλά έχουμε και συντονιστές των πολιτικών ομάδων από την Επιτροπή των Περιφερειών. Έχουμε τους κυρίους Αζοπάρντι, Πέτερσεν, Λόγκεν, Στένσον, Μπανάσακ, και οι καλεσμένοι αυτοί θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν το λόγο. Ας κανονίσουμε τη διαδικασία. Θα δώσω πρώτα το λόγο στον πρόεδρο της Επιτροπής ε, Φυσικών Πόρων της Επιτροπής των Περιφερειών, στον κύριο Μαρτικάινεν, για μια σύντομη παρέμβαση. Και κατόπιν θα δώσω το λόγο στον εισηγητή της ε, Επιτροπής Περιφερειών, στον κύριο Κιγιόμ Κρός, για, 10 λεπτά και κατόπιν θα ακούσουμε για δύο λεπτά τους ε, συντονιστές της Επιτροπής Γεωργίας και μετά τους συντονιστές από την Επιτροπή Φυσικών Πόρων της Επιτροπής των Περιφερειών. Ε, παρακαλώ να κοιτάτε το χέρι μου και το σφυράκι, γιατί μετά τα δύο λεπτά θα αρχίσω να το κουνάω επίμονα. Παρακαλώ κύριε Μαρτικά, να έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητά μέλη του Ευρωκοινοβουλίου, Κοινοβουλίου, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίε και κύριοι. Εξ ονόματο ε, τη Επιτροπή ΝΑΤ, τη Επιτροπή των ε, Περιφερειών, θα ήθελα να σα ευχαριστήσω που μα έχετε προσκαλέσει για δεύτερη συνεχή χρονιά στι συνεδριάσει τη Επιτροπή σα. Αυτή τη φορά θα συζητήσουμε το μέλλον τη κοινή γεωργική Πολιτική που θα είναι ένα από τα μείζωνα ζητήματα συζήτηση φέτος σε ευρωπαϊκό επίπεδο στο πλαίσιο τη ευρύτερη συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης και το μέλλον της ε, χρηματοδότησης στην Ευρώπη. Θα ήθελα να ακούσω και τις δικές σας απόψεις. Ε, όλοι μας εδώ, ε, μέλη της, της Επιτροπής αυτής, είμαστε πολιτικοί εκπροσώποι εκπρόσωποι των πολιτών. Είμαστε όμως και εμείς οι ίδιοι πολίτες ε, και προσπαθούμε να ανταποκριθούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις, ε, στα καθήκοντα που μας έχουν ε, εκχωρήσει οι ψηφοφόροι μας. Και εσείς βέβαια γνωρίζετε ποια είναι τα φλέγοντα ζητήματα σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Ωστόσο, είναι σημαντικό να ακούσουμε και τις απόψεις ε, των πολιτικών αυτών που δραστηριοποιούνται στις ε, πόλεις, στα χωριά, στις περιφέρειες. Γι' αυτό είναι σημαντική η σημερινή συζήτηση. Εν γέννη, η Ευρωπαϊκή Ένωση έρχεται αντιμέτωπη με μία σειρά προκλήσει, για παράδειγμα το Brexit και οι επιπτώσει ε, στον ευρωπαϊκό προπολογισμό, αυξανόμενο ευρωσκεπτικισμό και παγκόσμιε προκλήσει όπω η κλιματική αλλαγή και οι ελλείψεις και άλλες περιβαλλοντικές προκλήσεις. Η κοινή γεωργική πολιτική υπερβαίνει τους ε, συγκεκριμένους ε, τομείς. Ε, η κοινή γεωργική πολιτική αφορά την ασφάλεια φωτιασμού στην Ευρώπη, την βιώσιμη παραγωγή τροφίμων, την απασχόληση και τις οικονομικές ευκαιρίες στην Ήπεθρο, αφορά την υγιεινή διατροφή, την βιοπικιλότητα και την κλιματική αλλαγή. Γνωρίζουμε όλοι τις συζητήσεις του παρελθόντος και πόσο δύσκολο είναι να διαμορφώσουμε την κοινή γεωργική πολιτική με έναν τρόπο που να ικανοποιεί τους πάντες. Πριν επισέλθουμε στις λεπτομέρειες της συζήτησης, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να δούμε την κοινή γεωργική πολιτική ως μία από τις ε, μείζονες πολιτικές ε, που ε, μας συνδέουν και έτσι θα επιτρέπουν και στις πόλεις και περιφερειές μας, στην ύπεθρό μας και στις χώρες μας να, παρέχει, να παρέχουν ένα καλό βιωτικό επίπεδο σε όλους τους πολίτες. Η ΚΑΠ αφορά λοιπόν τη γεωργία, αλλά αφορά και τις ε, περιοχές ε, αυτές τις ε, τις γεωργικές, ε, όσους ε, ε, εποφελούνται από τις επαγγελματικέ ευκαιρίες στην Ήπεθρο, όσους μένουν μακριά από τα αστικά κέντρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προσωπικά πιστεύω ότι αφορά για τη διατήρηση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς και του κοινωνικού μας μοντέλου στη γεωργία μας. δεν μπορούμε να πάμε πίσω στον χρόνο, έχουμε όμως υποχρέωση να βελτιώσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση για τους πολίτες μας, για όλους τους πολίτες βλέπουμε ότι η 7η έκθεση συνοχής ε, διαπιστώνει σημαντική ανισορροπία στην ανάπτυξη μεταξύ ε, αστικών ε, και μη αστικών περιοχών. αυξάνα το κίνδυνο της ανέχειας στην Ήπεθρο σε σχέση με τα αστικά κέντρα. Υπάρχει μια αίσθηση εγκατάλειψης στην Ήπεθρο με αυξανόμενο ευρωσκεπτικισμό και αντίστοιχη συμπεριφορά και στάση στι εκλογικέ αναμετρήσει. Παρότι η συνοχή λοιπόν είναι στόχο στην, στην θήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό τη δεν αποδίδει αρκετή προσοχή σε τέτοια ζητήματα σε ό,τι αφορά τις ε, περιοχέ τη υπαίθρου. Η σημερινή συζήτηση για την ΚΑΠ είναι σημαντική. Ταυτόχρονα θα ήθελα να τη συνδέσω και με τη συζήτηση για το μέλλον τη Ευρώπη, Γιατί δεν εξετάζουμε μόνο έναν κλάδο της οικονομίας μας. Η γεωργία δεν είναι απλώς ένας, άλλος, ένας ακόμα κλάδος. Είναι η βάση της ύπαρξής μας και η Ευρώπη θα πρέπει να ε, το, την εξετάσει με την αντίστοιχη σοβαρότητα. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε κύριε Ματικά. Να δώσω τώρα το λόγο στον εισηγητή. Τον κύριο Κιγιόμ Κρός, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι βουλευτές, ο συγγετής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, της ΟΚΕ για την προοπτική 2020, θα ήθελα να αναφερθώ στις προτάσεις μας, στις συστάσεις μας για τις τοπικές και περιφερειακές προοπτικές της μελλοντική ΚΑΠ. ή ε, μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, που έχουν μπροστά μας, μας υποχρεώνουν να αναδιατυπώσουμε τους όρους της ΚΑΠ για να καταστεί μια πολιτική δίκαιη, βιώσιμη και αλληλέγγυη στην υπηρεσία του Γεωργού, της, ε, ε, των εδαφών, του καταναλωτή και του πολίτη χωρίς οικονομική, κοινωνική, περιβαλλοντική, εδαφική και διεθνή νομοποίηση η ΚΑΠ δεν μπορεί να επιβιώσει. Τι διαπιστώνουμε λοιπόν σήμερα, πλην όμως, ότι πολλοί είναι οι γεωργοί μεγάλο ποσοστό που έχουν είτε ανάξιο του μόχθου τους εισόδημα είτε πολλούν τα προϊόντα τους με ζημία. Ότι οι άμεσες πληρωμές είναι πολύ άνισα κατανεμημένες μεταξύ των εκμεταλλεύσεων και των κρατών μελών. Η βιοποικιλότητα, το κλίμα, το περιβάλλον, η δημόσια υγεία πληρώνουν βαρύτατο φόρο στην ε, επιλογή της υπερβολικά βιομηχανοποιημένης γεωργικής παραγωγής. Πολλές είναι οι περιοχές της υπαίθρου που χάνουν την ε, οικονομική τους ε, βάση επιβίωσης. είναι, πολλά είναι τα προϊόντα μας τα οποία εξάγονται σε τιμές χαμηλότερες ε, από το κόστος παραγωγής εις βάρος της επιβίωσης των γεωργών τρίτων. Ε, πρέπει λοιπόν να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες της γεωργίας. Είναι μεγάλη η πτυτικότητα των τιμών της γεωργίας. Είναι ασύμβατη με την επιβίωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και θεωρούμε ότι η ρύθμιση των αγορών για πολλούς τομείς της παραγωγής θα είναι πιο αποτελεσματική και λιγότερο δαπανηρή από ότι η ε, ανάπτυξη μέτρων εκ των υστέρων, ε, χωρίς λοιπόν ε, τιμές σωστές, γεωργικές τιμές, χωρίς οικονομική αναγνώριση. Ο νέος θα αποστρέψει το βλέμμα από το επάγγελμα του γεωργού ε, είναι μεγάλο, μεγάλη παγίδα η λύση της ε, εγγύησης ε, της ασφάλισης οδήματος, όπως άλλωστε αποδεικνύεται και από την εμπειρία των Ηνωμένων Εθνών. Έγινε η παρουσίαση της δουλειάς της Επιτροπής σας, του κανονισμού Omnibus και των λύσεων που θεωρούνται ωστόσο πολύ σημαντικές για το μέλλον της ε, ΚΑΠ ε, και εάν χάρη στη δουλειά σας μπορεί να δώσει περισσότερη δουλειά στο γεωργό ε, η γεωργία με μια πιο ευέλικτη και ομοιόμορφη εφαρμογή των κανόνων της γεωργίας, της κοινής γεωργίας στην Ένωση δεν θα μπορέσει παρόλα αυτά να λύσει τα προβλήματα της κρίσης. Γι' αυτό χρειάζεται μια διαφορετική προσέγγιση και συμμετοχή όλων των παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων και των καταναλωτών στις επιλογές, τροποποίηση ακόμα και του δικαίου του ανταγωνισμού, εάν καταστεί αυτό απαραίτητο. Περιμένουμε με ανυπομονησία τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο τομέα αυτό, γιατί τα στοιχεία της διάσκεψης για τις προοπτικές ε, στην οποία αναφέρθηκαν νωρίτερα το Δεκέμβριο, που έγινε το Δεκέμβριο είναι πολύ ανησυχητικά. Το, 70, το 60% της διάθεσης των γεωργικών προϊόντων το έχουν 7 παραγωγή και 5 με τα ε, ε, βιομηχανίες επεξεργασίας έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό των προϊόντων σε ε, το 56% της παραγωγής σε 13 κρατη το 2012. Έτσι λοιπόν περιμένουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να στηρίξει με όλο της το ειδικό βάρος την παραγωγή των ε, τροφίμων, μια τροποποίηση όπως θα πρέπει να γίνει γιατί είναι αρκετά απαρχαιωμένοι αυτοί οι κανόνες από το 1994 προκειμένου να προχωρήσουμε σε νέες εμπορικές σχέσεις και περιμένουμε να δούμε με τη διάσκεψη 8ης Μαρτίου πώς μπορούμε να τροποποιήσουμε τους σχετικούς κανόνες. Οι άμεσες ενισχύσεις ανά εκτάριο θα πρέπει να βρουν ένα ανώτατο επίπεδο και μια διαρρύθμιση ανάλογα με τη γεωργική εκμετάλλευση για να γίνει η μια ζώσα ύπεθρος, για να έχει την ευκαιρία και ο νέος γεωργός, γιατί η μεγάλη βιομηχανική εκμετάλλευση δεν είναι δυνατόν να εκχωρηθεί. Το ε, ανώτατο όριο σε 60 με 100.000 ευρώ σε άμεσε ενισχύσει ανεκμετάλλευση δυστυχώ δεν αναφέρεται παρότι είναι απαραίτητο για μια δίκαιη ΚΑΠ στην ανακοίνωση για την ΚΑΠ 2020 που παρουσίασε στι 29 Νοεμβρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρέπει οπωσδήποτε να μεριμνήσουμε για τα 10 εκατομμύρια γεωργικών εργαζομένων ε, που πολλές φορές ε, εργάζονται σε μερική απασχόληση για μισθούς πείνας και πολλές φορές και παράνομα. Ζητούμε να γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα των, ε, εργατών, των εργαζομένων στη γεωργία, να μειωθούν οι άμεσες ενισχύσεις ε, και να μην χορηγούνται αυτές όταν μια ε, γεωργική εκμετάλλευση δεν τηρεί τις κοινωνικές προδιαγραφές που ισχύουν στη χώρα μέλος. Επίσης θα πρέπει να επιμείνω ως προς την αναγκαιότητα για μεγαλύτερη επαγρύμψη σε σχέση με την υπερβολική αυτοματοποίηση των γεωργικών τεχνολογιών και την όλο και μεγαλύτερη παρέμβαση του big data των μεγάλων ε, όγκων δεδομένων. Θα πρέπει να μην ξεφύγει από τον έλεγχο του γεωργού η εκμετάλλευση, να έχει αυτό την αυτονομία της απόφασης και θέλουμε βέβαια πρασίνισμα που θα συνοδεύει, θα παρακολουθεί παρακολουθεί το γεωργό στη μετάβαση προς ε, ε, τρόπους παραγωγής που θα είναι πιο ευνοϊκοί για το περιβάλλον, για τη βιοπικιλότητα και το κλίμα, η εναλλαγή των ε, η αμυψισπορά, η διατήρηση μόνιμων χορτολιβαδικών εκτάσεων, η αποφυγή των χημικών στην παραγωγή κτλ. Θέλουμε τιμές πολύ πιο δίκες και με το το επίπεδο στήσαμε σε ε, με ένα με μια οροφή στι άμεσε ενισχύσει μπορούμε να κάνουμε οικονομία σε άλλου τομεί, από τον πρώτο τομέα που μπορεί να μα επιτρέψει να εξισορροπήσουμε το δεύτερο τομέα για μια βιώσιμη ανάπτυξη. Από τι προτεραιότητε του δεύτερου ε, πυλώνα θα ήθελα να υπογραμμίσω την υποστήριξη στι σύντομε αλυσίδε διάθεση των προϊόντων, την υποστήριξη στη τεχνολογική καινοτομία και την κοινωνική ε, καινοτομία για του ε, τρόπου παραγωγή, μετατροπή μεταποίηση και διάθεση που θα είναι βιώσιμη υποστήριξη στην ε, συλλογική εστίαση, ε, σημεία ένταξης ε, για όλες τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την Ήπεθρο, η ικανοποίηση των αναγκών της Ήπεθρου που δεν εξαντλούνται σε αυτά που μπορεί να προσφέρει η ΚΑΠ και η, περιφερεια, η ανάπτυξη της Ήπεθρου, η μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών για σε σχέση με τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό που αφορά τις ζώνες της υπαίθρου αποδεικνύει ότι αυτό είναι ανεπαρκή σε σχέση με τη σημασία αυτών των ζώνων στην Ευρώπη. Χρειάζεται λοιπόν μια επανεξορρόπηση του προϋπολογισμού στα διαρθρωτικά ταμεία των οποίων η συνεισφορά στην ανάπτυξη υπαίθρου έχει μειωθεί σημαντικά ενώ και μεγαλύτερη συνεργασία θα απαιτηθεί και συνδυαστική δράση και απλοποίηση ενεργοποίηση ταυτόχρονα των πόρων των διαφόρων ευρωπαϊκών ταμείων καθώ και η υιοθέτηση μια ημερήσια ημερήσιας ενό θεματολογίου για την Ήπεθρο. Για να ολοκληρώσω λοιπόν κάνουμε τώρα το σχεδιασμό τη Ευρώπη και του μέλλοντό τη. Η ε, οικοδόμηση μια δίκαιη, βιώσιμη και αλληλέγγυα ΚΑΠ δεν μπορεί παρά μόνο να γίνει μέσα σε μια Ευρώπη δίκαιη, βιώσιμη και αλληλέγγυη. Δεν μπορούμε παρά να κάνουμε τι σωστέ επιλογέ και σα ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίαση ε, μετά την ανακοίνωση και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την νέα προσέγγιση που συνδέεται και με την προετοιμασία των στόχων και των αξιών ε, που ετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και που θα χαρακτηρίσουν την μελλοντική και σημαντικό ρόλο θα διαδραματίσουν και οι περιφέρειες και καλό θα είναι λοιπόν οι περιφέρειες να καταθέσουν τι δικέ τους προτάσεις. Γιατί είναι πολύ διαφοροποιημένη η Ευρωπαϊκή Γεωργία, οι αρχές, οι αξίες και οι στόχοι τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αξιοποιώντας όμω το ιδιαίτερο δυναμικό κάθε μεμονωμένης περιφέρειας. Γιατί και θεματικέ ε, διαφοροποιήσει υπάρχουν, αλλά και πολλέ περιφερειακέ ιδιαιτερότητε. Όλα αυτά τα επιμέρου στοιχεία είναι σημαντικό να τα αξιοποιήσουμε περιφερειακή πραγματικότητα. Θα δώσω τώρα το λόγο πρώτα στην κυρία Μίλλερ. Η Επιτροπή των Περιφερειών έρχεται να συζητήσει μαζί μας και στις όλες αυτές οι βοήθειες, οι οικογένειες οι οποίες διαχειρίζονται μικρές μεσές εκμεταλλεύσεις πρέπει να ενισχυθούν βεβαίως ε, με ό,τι σχόλια έχετε να μας προσφέρετε για να βελτιωθεί η δυνατότητα επιβίωσης και προσανατολισμού προς το μέλλον των ε, γεωργικών εκμεταλλεύσεων και είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι έχουμε αυτές τις δύο συζητήσεις για την κοινή γεωργική πολιτική σε πρώτο στάδιο με μέλημα την παραγωγή υγιών γεωργικών προϊόντων και τροφίμων. Και έτσι, ορισμένες φορές, η Ευρώπη σε αυτό δεν ήταν πάντα επιτυχημένη. Το στο δημοσιονομικό πλαίσιο αναφέρθηκε. Νομίζω ότι μπορούμε εδώ από το Κοινοβούλιο να συμβάλλουμε στη διαμόρφωση και ε, λύσεων. Ε, ασφαλώς το γεγονό ότι περικόπτονται τα κονδύλια για τη γεωργία δεν μας χαροποιεί. Μάλλον θα έπρεπε να ενισχυθούν, μάλλον θα έπρεπε να αναπτυχθεί η πολιτική της συνοχής. Είμαστε πεπισμένοι ότι διακυβεύονται πολύ περισσότερα από την ε, η γεωργική εκμετάλλευση, το οδήποτε τρόφιμο που παράγεται στην Ευρώπη. δεν έχουμε να κάνουμε με την ενίσχυση και διατήρηση της υπαίθρου με την ενότητα, με την κοινωνική συνοχή, με τις λιγότερο ισχυρές περιφέρειες, με τον, με τον ανθρώπινο παράγοντα και την επαφή των ανθρώπων μέσα από τα χωριά, μέσα στα χωριά, γιατί στις πόλεις το ίδιο δεν συμβαίνει. Η γεωργική πολιτική βεβαίως βρίσκεται ενώπιον τεράστιων προκλήσεων. Χαίρομαι που έχουμε την ευκαιρία να συνεργαστούμε εδώ και προκλήσεις ένταση εργασίας οπωσδήποτε. Η Ήπεθρος θα πρέπει να βρεθεί στο επίκεντρο των μελημάτων μας, ναι. Η γεωργία. Έχουν μειωθεί κατά 40% τουλάχιστον οι γεωργοί κτηνοτρόφοι που παράγουν ε, γάλα. Πρέπει λοιπόν ε, πάνω απ' όλα να στρέψουμε το βλέμμα στον γεωργό και ακτινοτρόφο. Επίσης το θέμα του περιβάλλοντος πρέπει να μας απασχολήσει με δύο μεγάλους χαμένους εδώ από τη γεωργική πολιτική. Η βιοπικιλότητα δηλαδή όσο πιο εντατική είναι η γεωργική εκμετάλλευση, η βιομηχανική γεωργική εκμετάλλευση χάνεται βιοπικιλότητα και δεν μπορούμε αυτό να το να το λησμονήσουμε, να το αποκρύψουμε ή να το παραμελήσουμε. Είναι κάτι που πρέπει να απασχολεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ε, ακούστηκαν διάφορες ε, ιδέες ε, γενικά, γενικές, αφηρημένες ως από απλοποίηση κτλ. Τι ακριβώς όμως αυτό συνεπάγεται, κύριε Χόμπεν, δεν, δεν το ξέρει κανείς. Περιμένουμε να δούμε συγκεκριμένες προτάσεις. Αυτό που δεν θα θέλαμε όμως θα ήταν στο τέλος να αυξηθούν όλο και περισσότερο οι αποκλήσεις να μειωθεί η συνοχή στη γεωργία στην Ευρώπη, να περάσουμε σε μια επανεθνικοποίηση. Αυτό θα ήταν τεράστιο λάθο. Θα ήταν μια τεράστια απώλεια σε σχέση με ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, μια κοινή ανάπτυξη στη γεωργική πολιτική, η οποία βεβαίω θα πρέπει να συνεχίσει, πάντα με διατήρηση βεβαίω ενό σε περιφερειακό επίπεδο ε, περιθωρίου ε, χειρισμών ή διακριτική ευχέρεια. Ε, Επίση, για το θέμα τη ε, θέσεως της γεωργίας στις εμπορικές αλυσίδες. Είναι κάτι το οποίο πρέπει στην ε, ε, αλυσίδα δηλαδή της, του εμπορίου των προϊόντων. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε θεωρητικά μόνο να συζητούμε πως κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η κατάσταση επιδεινώνεται. Βλέπουμε ποια είναι η κατάσταση σε άλλα κράτη, εξαγωγές και όλα αυτά. Δυστυχώς εμείς βρισκόμαστε ακόμη σε επίπεδο συζήτησης ότι υπάρχουν κακές δομές στην Ευρώπη. Αυτό εμείς στην Ευρώπη έχουμε πολύ διαφοροποιημένη γεωργία που δεν περιορίζεται στον γεωργικό προϋπολογισμό. Έχουμε και την ενιαία εσωτερική αγορά και θα πρέπει στους μηχανισμούς που έχουμε να λάβουμε υπόψη τις ιδιαιτερότητες των περιφερειών στην κοινή γεωργική μας πολιτική. Ακόμη και εντό της ίδια περιφέρειας υπάρχουν διαφοροποιήσεις πολλές φορές στην Ευρώπη. Συγγνώμη που χρειάστηκε να το τονίσω, αλλά θεωρώ ότι είναι το κλειδί στην όλη συζήτηση άλλο η γαλακτοπαραγωγή στη Φιλανδία και άλλο η γαλακτοπαραγωγή στη Γαλλία ή την Πολωνία. Μεγάλη διαφοροποίηση υπάρχει. Με προβλημάτισε αυτό το έγγραφο, γιατί μπορεί κανείς να πιστεύει σε έναν φανταστικό κόσμο όπου όλα βαίνουν καλώς, αλλά εδώ θέλουμε και επιδοτήσεις προς τους γεωργούς ε, και προσαρμοσμένες ε, στο, στην εργασία. Πολύ καλά ακούγονται όλα αυτά, αλλά πώς ακριβώς ε, θα τα ορίσουμε όλα αυτά. Γιατί μπορεί να πει ο Γιώργο ότι και τα πέντε μου παιδιά είναι γεωργική ε, εργασία. Πολύ καλά ακούγονται όλα αυτά, αλλά πώ ακριβώ ε, θα τα ορίσουμε όλα αυτά. Γιατί μπορεί να πει ο Γιώργο ότι και τα πέντε μου παιδιά είναι γεωργική ε, εργασία. υπό τον πυλώνα 1 σε αυτή τη βάση. Είναι ένα γραφειοκρατικό εφιάλτη και ελπίζω να μην ακολουθήσουν αυτή την άγουσα. Μια άλλη ώρα. Από την άλλη, από να του λένε ότι όχι δεν θα αξιοποιηθούν στην αγορά, θα πάρουμε προϊόντα από άλλες ε, χώρες που... Ο κύριος ähm, Έχοντας μελετήσει το έγγραφο, θέλω να ευχαριστήσω την Επιτροπή των Περιφερειών και προσφοράς. Πιστεύουμε εμείς ότι χρήμα δημόσιο πρέπει να χορηγείται μόνο εκεί όπου υπάρχει δημόσια προσφορά, προσφορά στο, ε, στην κοινή ε, προσφοράς. Πιστεύουμε εμείς ότι χρήμα δημόσιο πρέπει να χορηγείται μόνο εκεί όπου υπάρχει δημόσια προσφορά, προσφορά στο, ε, στην κοινή ε, για να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή και από την άλλη ταυτόχρονα με άλλα κονδύλια του προπολογισμού να ενισχύουμε πολιτικές οι οποίες επιδεινώνουν τι κλιματικέ συνθήκε. Επίση, στη χρήση των ζυζανιοκτώνων για τα οποία έγινε λόγος υπάρχει μια τελευταία μελέτη ε, στη Γερμανία που δείχνει ότι τα πτερωτά έντομα έχουν μειώσει. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Αζοπάρντι. Μετά το 2020 θα πρέπει πρώτα απ' όλα να ενισχύσει τη θέση των γεωργών στην αγορά για να αποτρέψουμε την, το κλείσιμο των γεωργικών τα κονδύλια του, των γεωργικών ταμείων εις βάρος των άμεσων ενισχύσεων. Θα πρέπει να ισχύει μεγαλύτερη επικουρικότητα για τη μεταφορά κονδυλίων από τα κράτη-μέλη από τον πρώτο στο δεύτερο σε ιδιωτικά μέσα για να, να αποτρέψουμε τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές και τη μεγάλη αστάθεια των τιμών. Μόνο έτσι θα κάνουμε ελκυστική την γεωργία, θα είναι γάλακτος και βουνά βουτύρου. Θα πρέπει να γίνει σωστός ε, σχεδιασμός γιατί η υπερβολική γραφειοκρατία θα έχει τα αντίθετα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Επίση, θα ήθελα συμφωνίε ελεύθερου εμπορίου που συνάπτουμε με τρίτε χώρε. Σα ευχαριστώ για την προσοχή σα και προσβλέπω σε συνέχιση τη αγαστή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Ο κύριο ε, Ούνοβρε. Νομίζω ότι είναι απαραίτητο τι προκλήσει που αντιμετωπίζει η κοινωνία. Η απορρίθμιση ευνόησε τη συγκέντρωση της παραγωγής ε, στις περιφέρειες έντασης εργασίας με, ε, για τα μέτρα οικολογικοποίησης. Χρειαζόμαστε μια ρηξικέλευτη μεταρρύθμιση της κοινή γεωρικής πολιτικής. Μια αναθεώρηση της κάπου που θα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια βιώσιμη γεωργία με φιλοπεριβαλλοντικές ε, και φιλοκλιματικές πρακτικές. Επίσης θα πρέπει να δώσουμε έμφαση στον τοπικό και περιφερειακό παράγοντα και τις πρακτικές. Ε, αυτές είναι ε, και οι προτάσεις της Επιτροπής ε, της Γεωργίας. Θέλουμε μεγαλύτερη εγκύτητα, μεγαλύτερη περιφερειακή ανάμεξη, γιατί τα μέτρα θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την τοπική, κοινωνικο-οικονομική και περιβαλλοντική πραγματικότητα. Και γι' αυτό θα πρέπει και οι οι ΟΤΑ που καλούνται να εφαρμόσουν αυτά τα μέτρα να συμμετέχουν και στο σχεδιασμό τους. Επίσης, ο καταναλωτής γίνεται όλο και πιο απαιτητικός απαιτεί υγιεινά, τοπικά, βιολογικά προϊόντα. Ο καταναλωτής θέλει να γνωρίζει τι βάζει στο στόμα του. Ε, και γι' αυτό μόνο με μια ισχυρή κοινή γεωρική πολιτική θα εξασφαλίσουμε πραγματική επιστημιστική ασφάλεια για τον καταναλωτή. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρίες και κύριοι. Η προσπάθεια και το διακύβευμα της κοινή γεωργικής πολιτικής δεν μπορεί πλέον να συνεχιστεί για να, και να πληρεί τη βελτίωση της κλιματικής αλλαγής. Θα πρέπει όλα αυτά να προστεθούν. Δεύτερον, πρέπει να υπάρχει ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολλές από τις προκλήσεις όπως ε, εντό ε, του γεωργικού κλάδου. Όμω η ε, μετάβαση αυτή είναι αργή και απαιτεί περισσότερε επενδύσει σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη καινοτομιών. Η κοινή γεωργική πολιτική λοιπόν, ε, ε, ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού και ε, ένας σωστός προπολογισμό είναι απαραίτητα στοιχεία. Τέλος, θα πρέπει να είναι πιο απλή η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για επιδοτήσεις. Αυτή τη στιγμή υπάρχει διοικητικό άχθος και μεγάλο ρίσκο και, είναι, κακή, κακές, είναι δύσκολη η πρόσβαση στα χρηματοδοτικά εργαλεία για τις μικρές επιχειρήσεις και έτσι μένουν πίσω. Σας ευχαριστώ κύριο Στένσον. Εγώ ε, συνέταξα και έκθεση πρωτοβουλία για την ανανέωση τη υπαίθρου και για τα έξυπνα χωριά σχέση με τα αστικά κέντρα, τι αστικέ περιοχέ. Και αυτό εν μέρει οφείλεται στην ανάπτυξη των μεγάλων αστικών κέντρων και των πρωτευουσών που καταλαμβάνουν όλο και μεγαλύτερο χώρο ενώ η Ήπεθρος πασχίζει για να εξασφαλίσει ε, ευκαιρίες, υποδομές και απασχόληση στους νέους και να προσελκύσει εργαζομένους. Ενώ ε, έχουμε την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για, τη, για τα ευρωπαϊκά χωριά, ε, έξυπνα χωριά. Θα πρέπει έτσι να στηρίξουμε την Ήπεθρο για να γίνει βιώσιμη η Ήπεθρο. Δεν αρκεί όμως η πρωτοβουλία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Λυπάμαι για την έλλειψη φιλοδοξία που επέδειξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί αξιοποιεί προηγούμενε πρωτοβουλίε θα περιληφθούν και αυτές στο θεματολόγιο για την Ήπεθρο. Και λυπάμαι που η διακήρυξη Κάρσα, ε, του ΚΟΡΚ δεν ε, ε, υλοποίησε τους στόχους και έμεινε στα χαρτιά. Θα πρέπει ε, μια δεύτερη διακήρυξη του ΚΟΡΚ να μην παραμείνει στη θεωρία και απλώς στα χαρτιά. Θα πρέπει να ε, τις δώσουμε σάρκα και οστά ότι συμμετέχουμε σε μια σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει η ίδια ευρυζωνικότητα στι τηλεπικοινωνίε να εξασφαλίζεται παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι σε μερικά μόνο σημεία ότι συμμετέχουμε σε μια σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει η ίδια ευρυζωνικότητα στι τηλεπικοινωνίε να εξασφαλίζεται παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι σε μερικά μόνο σημεία. Επίση, θα πρέπει να έχουμε ευρυζωνικό Ιντερνετ υψηλή ταχύτητα και στην Ήπεθρο και να μην περιορίζουμε την πρόσβασή του σε ορισμένα κρατημέλη ανάλογα με τι επενδύσει που κάνουν στην ευρυζωνικότητα. Επίση, θα πρέπει να έχουμε πρόσβαση σε επενδύσει για σχέδια ευρυζωνικότητα και μεγάλη εμβέλεια και να βελτιώσουμε την κατάσταση, να δημιουργήσουμε αντιπαράθεση μεταξύ αστικών και ε, μη αστικών περιοχών, αστικών περιοχών και υπαίθρου. Θα πρέπει να αλληλοστηρίζονται και να αλληλοβοηθούνται τα αστικά κέντρα με την υπαίθρο. Ε, μόνο έτσι θα κρατήσουμε τον αγροτικό πληθυσμό στην Ήπεθρο. Να μην περιορίσουμε μόνο ως μονόδρομο με βάση την πρωτοβουλία του ΚΟΡΚ. Θα πρέπει να, να εξασφαλίσουμε τη συμμετοχή των ΟΤΑ για να αξιοποιήσουμε στο έπακρο το δυναμικό της Ήπεθρου είτε με γραφεία που θα προωθούν τις επιχειρήσεις, θα τους βοηθούν στην υποβολή προγραμμάτων για διαγωνισμούς και το καθεξής. Επόψε μπορούμε να προωθήσουμε αυτό το θεματολόγιο προς όφελος όλων των αγροτικών περιοχών και ελπίζω αυτό να γίνει όσο το δυνατόν συντομότερα γίνεται. Σας ευχαριστώ. κύριο κύριος Άνταμ Μπανάσακ. Αξιότιμη Ευρωβουλευτέ, ε, ε, αγαπητοί συνάδελφοι από την Επιτροπή Περιφερειών και την ΕΟΚΕ. Εκ μέρους της ε, ομάδας ε, συντηρητικών και μεταρρυθμιστών της Επιτροπής Περιφερειών θα ήθελα να σας ευχηθώ καλή χρονιά και να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον πρόεδρο της Επιτροπής Γεωργίας γιατί ότι απαιτούμε μεγαλύτερη ελαστικότητα στην άσκηση της κοινή γεωργικής πολιτικής. Πολύ σωστά στην ανακοίνωσή της η η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει ότι είναι υπερβολικά διεξοδικέ οι διατάξει και λεπτομεριακέ και δεν, λαμβάνουν, δεν εφαρμόζονται λαμβάνοντα υπόψη τι περιφερειακέ ιδιαιτερότητε. Γι' αυτό χρειάζεται μεγαλύτερη ευελιξία. Γιατί οι ιδιαιτερότητε ε, είναι κυρίω περιφερειακέ σε ό,τι αφορά τη γεωργία. Γι' αυτό και η ευρωπαϊκή γεωργική, κυρία γεωργική πολιτική θα πρέπει με ελαστικότητα να εφαρμόζεται. Είναι σημαντικό για την υλοποίηση των εθνικών στόχων. Δεν θα πρέπει να μα υπαγορεύουν οι Βρυξέλλε του ε, ε, στόχου κεντρικά. Επίσης, ε, σίγουρα θα πρέπει να διαφυλάξουμε την, πολιτική, την γεωργική πολιτική με τους δύο πυλώνες θα να δίνεται τέτοια δυνατότητα μεταφορά κονδυλίων μεταξύ των δύο πυλώνων από τα κράτη-μέλη. Επίση, απευθύνω έκκληση να μην περιπλέξουμε, να μην δυσχεράνουμε την κοινή γεωργική πολιτική. Όσο πιο απλή είναι, τόσο πιο εύκολα θα εφαρμόζεται. Γιατί σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο πολύ συχνά αντιμετωπίζουμε προβλήματα με τι γραφειοκρατικέ και περίπλοκε διατάξει. Θα πρέπει να αφήσουμε. Σα ευχαριστούμε, κύριε Μπανάσακ. Πιο αυστηρό στην τήρηση του χρόνου. Κύριο Ροπέ, πρώτα, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι μα από την Επιτροπή των Περιφερειών. Και εγώ υπήρξα Δήμαρχο για μεγάλο χρονικό διάστημα και με ενδιαφέρουν ιδιαίτερα οι δραστηριότητε σα. Σα ευχαριστώ λοιπόν πολύ που ήρθατε και μας παρουσιάσατε τις απόψει και προτάσεις σας. Βλέπω ότι συμφωνούμε σε πολλά σημεία. Το ερώτημα είναι, συμπεριλαμβάνει όλους ε, τους στόχους μας. Πολύ σωστά λέτε ότι η νεολαία εγκαταλείπει τη γεωργία. Αυτό συζητήσαμε και νωρίτερα σήμερα. Μάλλον όλοι ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε, αλλά πρέπει να αρχίσουμε από τώρα για να διαμορφώσουμε την περίοδο μετά το 2020. Τα κράτη-μέλη έχουν πάνω από το 50% της πρωτοβουλίας ε, λήψης υποφάσεων για τις ε, γεωργικές επιδοτήσεις. Οπότε είναι και αυτό ένα σημαντικό στοιχείο γιατί υπάρχει σημαντική ανισομέρεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν αποδίδεται παρκής προσοχή στις περιφέρειες ε, που υστερούν. Και συμφωνώ ότι η αξία των στοιχείων είναι πολύ χαμηλότερη σε αυτές τις περιφέρειες και ουσιαστικά φυτοζωούν αυτές τις περιοχές. Και ελπίζω οι αποφάσεις να ε, βοηθήσουν αυτές τις περιοχές. Και θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη συνεργασία στον γεωργικό τομέα. Ένα από τα σημαντικά ζητήματα είναι μια δίκαιη αλυσίδα πληρωμών. Πολύ συχνά ο γεωργικός τομέας παίρνει μόνο τα υπολείμματα. Είναι τόσο χαμηλές ε, οι επιδοτήσεις ε, και οι πληρωμές που μπορεί απλώς να επιβιώσει, αλλά όχι να ευημερήσει ο κλάδος. Θα πρέπει ε, η περιφέρεια των Γιώργο. Είναι πολύ σημαντικά αυτά τα στοιχεία. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η ανταλλαγή απόψεων. Τα μέλη της Επιτροπής των Περιφερειών έχουν να μας ε, εκπροσωπούν εδώ τις ε, θέσεις των περιφερειών, των τοπικών αρχών, αλλά βέβαια και καθώς είναι πολύ κοντά στον Γεωργό έχουν τις Ευρωπαϊκές Ένωση η Γεωργία. Να, μην, να είναι δηλαδή η Γεωργία η πολιτική αυτή στην οποία μόνο χαμένοι υπάρχουν. Δεν πρέπει να το βλέπουμε έτσι. Υπάρχουν πολλοί γεωργοί στην Ευρώπη οι οποίοι μια χαρά τα βγάζουν πέρα, κερδίζουν χρήματα. Και αν δεν συνέβαινε αυτό, τα 55 χρόνια ιστορίας που έχει πίσω της η ευρωπαϊκή κοινή γεωργική πολιτική θα ήταν ε, ε, μια μεγάλη αποτυχία νομίζω ότι καλό θα ήταν να στηριχθούμε σε αυτά που έχουμε, να μην προσπαθήσουμε δηλαδή να ανακαλύψουμε ή να εφεύρουμε καλύτερα από την αρχή τα πάντα. Στον πρώτο πυλώνα έχουμε στοιχεία που μπορούν να μας βοηθήσουν, ενισχύουν τη γεωργική οικογένεια, τη μικρή εκμετάλλευση, αν κοιτάξουμε τα τελευταία χρόνια και κυρίως τις επενδύσεις από τα μεγάλα ταμεία στην ΕΠΕ, συνάδελφων από την Επιτροπή των Περιφερειών. Ασφαλώς χρειάζεται ένας ισχυρός δεύτερος πυλώνας, χρειάζεται δηλαδή καλή οργάνωση της υπαίθρου που θα είναι και μόνο εάν βλέπει και καλές προοπτικές αλλά και τη δυνατότητα για ε, καλή γεωργική δραστηριότητα μπορεί να αποφασίσει ο νεαρός ε, να εγκατασταθεί ως γεωργός. Αυτό και για να ολοκληρώσω, ε, ο δεύτερος πυλώνας έχει λιγότερο. Πόσα από, τη δεύτερη, από το δεύτερο πυλώνα αντίστοιχα και ίσως έτσι μπορούμε να κάνουμε μία σύγκριση. η οποία θα η οποία θα καθιστά τα πράγματα και τις διαφορές πιο ορατές. Ευχαριστώ πολύ, κύριος Αντριού. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την... Ασχολούμαστε πολύ με το νέο πρότυπο που θα έχει μεταρρυθμίσει και πολύ σωστά ε, θέσατε και πολύ εύστοχα τα ζητήματα εν ώψη της μεταρρύθμισης. Σήμερα η ΚΑΠ δεν να καινοτομήσουμε σήμερα. Το επισήμαναν πολύ. Επίσης θα πρέπει να ξεκινήσουμε κατά τη γνώμη μου μια μεταρρύθμιση ε, τολμήρη στην κυνηγιορική πολιτική ειδικά για την περίοδο μετά το 2020 μέχρι το 2026. Επίσης, κάνατε το σύνδεσμο που το επισημάνατε, είναι το πώς θα εξασφαλίσουμε το γεωρικό εισόδημα, πώς θα εγγυηθούμε το γεωρικό εισόδημα και κυρίως ε, το εισόδημα των νέων ε, αγροτών. Γιατί δεν θα έχουμε βιωσιμότητα της γεωργίας αν δεν εξασφαλίσουμε το εισόδημα των ε, βασικών παραγόντων της γεωργίας, που είναι οι γεωργοί. Η μεταρρύθμιση δυστυχώ ε, ήταν αυτορυθμισμένη σε αγορέ, θα το είχαμε δει, αλλά από την πρόσφατη γαλακτοκομική κρίση διαπιστώσαμε ότι δεν επαρκούν οι αγορέ ε, ε, για να αυτορυθμιστούν. Χρειαζόμαστε κάποια μέσα ρύθμιση και εξασφάλιση. Επίση, αυτό ο ρυθμιστού. Χρειαζόμαστε κάποια μέσα ρύθμιση και εξασφάλιση. Επίσης, ε, αυτός ο κανονιστικός υπερθεματισμός δεν μας εξυπηρετεί. Θα πρέπει να ε, εξασφαλίσουμε ένα είδος κυκλικών συμβάσεων στη Γεωργία και να λάβουμε υπόψη τις προτάσεις σας, να εξασφαλίσουμε το γεωργικό εισόδημα στην Ήπεθρο, λαμβάνοντας υπόψη κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια και στη Γεωργία και να λάβουμε υπόψη τις προτάσεις σας, να εξασφαλίσουμε το γεωρικό εισόδημα στην Ήπεθρο, λαμβάνοντας υπόψη κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια και το ίντερνετ δεν έχει νοσοκομεία, δεν έχει υποδομές. Ευχαριστώ πολύ ενδιαφέρουσα η έκθεση. Ελληνικό Ιντερνετ δεν έχει νοσοκομεία, δεν έχει υποδομέ. Ευχαριστώ πολύ ενδιαφέρουσα η έκθεση. Το Κάποιοι λένε αν έφαγες κάτι σήμερα να ευχαριστήσεις τους ε, Γεωργούς. Όμως οι περισσότεροι έχουν, δεν είχε γίνει σωστά η σύγκληση, θα είχαν λάβει 11 εκατομμύρια παραπάνω το χρόνο. Πολύ ωφέλιμο, όχι μόνο για τα αστικά κέντρα, αλλά και για τους απλούς πολίτες και κατοίκους της υπαίθρου, τι τοπικές επιχειρήσει για όλους. Όμω, τι έγινε τελικά. Και εμεί πήραμε αυτή την απόφαση, στην Ιρλανδία, όχι στην Ευρώπη. Εγώ ε, Είμαι επικριτικό απέναντι στην Ευρώπη σε πολλά σημεία, αλλά πολλοί κοινότητε θα δώσαμε στο Λάρι Γκούντμαν και του φίλου του. Αν θέλουμε να αλλάξουμε τα πράγματα την επόμενη φορά, θα πρέπει να ε, λάβουμε μια πολιτική απόφαση. Ποιοι θα υποφεληθούν τελικά, αυτοί που παίρνουν το ιδιωτικό του αεροπλάνο για να ταξιδέψουν ή αυτοί που μοχθούν κάθε μέρα. Εγώ ξέρω με τι είναι το πλέον τα προβλήματά μα, γιατί η λύση βρίσκεται στα χέρια μα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ που μας δίνετε τη δυνατότητα και την ευκαιρία να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει συνεργασία μεταξύ των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Επιτροπή των Περιφερειών και ΕΟΚΕ. Έχουμε αυτά. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει συνεργασία μεταξύ των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Επιτροπή των Περιφερειών και ΕΟΚΕ. Έχουμε συναφείς ε, προτάσεις. Πρέπει να διασφαλίσουμε ένα καλύτερο βιωτικό επίπεδο στην Ήπεθρο. Αυτό αποτελεί ε, μείζωνα προτεραιότητα. Η γεωργική δραστηριότητα είναι πολύ σημαντική. Θέλουμε να υπάρχει ε, επιστηστική ασφάλεια και καλή. Αυτό ήδη περιλαμβάνεται στην κοινή γεωργική πολιτική, δεν χρειάζεται να τα ξαναπώ εγώ χρειαζόμαστε διαφορετικά, διαφορετικές λύσεις ανάλογα με το κάθε οικοσύστημα. Τι είναι σημαντικό τώρα, να διασφαλίσουμε επαρκή χρηματοδότηση ε, μέσω των ευρωπαϊκών κονδυλίων και σωστή κατανομή τους. Σε σωστή κατανομή ανάλογα και με το μέγεθος ε, του κάθε εμπορευμένου να υπάρχουν ίσες ευκαιρίες για όλους και πρέπει να δούμε πώς θα δημιουργηθεί μεγαλύτερο κέρδος στο πλαίσιο της ε, διατροφικής αλυσίδας. Αυτή η παραγωγή που, θα, ε, που παράγουν τα βασικά προϊόντα θα παράγουν όλα ένα και λιγότερο όσο περνάει ο καιρός λόγω των νέων τεχνολογιών. Χρειαζόμαστε λοιπόν βασικές υποδομές, ε, χρειαζόμαστε ευρυζωνικά δίκτυα, σύγχρονες προσεγγίσεις στην θέση σε εμπορία, σε ό,τι αφορά τώρα την ε, μεγαλύτερου τους μεγαλύτερους. ληστική προσέγγιση απαιτείται σε ό,τι αφορά την, ε, ανάπτυξη στις ε, τις διαφορετικές περιστάσεις σε κάθε χώρο. κύριος Νίκολσον, ευχαριστώ πολύ. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη της Επιτροπής των Περιφερειών για μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση, την οποία μελέτησα με μεγάλο ενδιαφέρον σε ό,τι αφορά την ισορροπία, για παράδειγμα, μεταξύ αστικών και μη αστικών περιοχών, αλλά ε, ρεαλιστικά μπορούμε να πούμε ότι και εντός των αστικών κέντρων υπάρχει μεγάλη ενισομέρεια, οπότε δεν υπάρχουν ουσιαστικά λύσει. Είναι ένα ευχολόγιο περισσότερο, χωρί να θέλω να σας επικράνω. Μου θυμίζει ε, τις ημέρες της ε, παλιότερα που δεν, υπήρχαμε, ε, που δεν υπήρχε η συναπόφαση και απλώς κάναμε λίστες με όλα αυτά που θα θέλαμε να πετύχουμε, αλλά τίποτα από όλα αυτά δεν ήταν εφικτό. Νωρίτερα κάναμε μια συζήτηση για το κατά πόσο ε, η γεωργία είναι ένα απλό επάγγελμα ή κάτι παραπάνω. Η αλήθεια είναι ότι αν δεν έχουμε γεωργική βιομηχανία που να είναι αξιόπιστη, ε, και αποδοτική κερδοφόρος, τότε ε, θα συνεχιστεί αυτή η τάση από τις γεωργικές περιοχές προς τις αστικές. Φεύγουν λοιπόν οι άνθρωποι από την Ήπεθρο γιατί θέλουν να βελτιώσουν το βιωτικό τους επίπεδο. Αυτό συμβαίνει στην πράξη. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Και θα έχουμε ακόμα μια συζήτηση στις 2 το μεσημέρι σήμερα για να εξετάσουμε το μέλλον της κοινή γεωργικής πολιτικής και το βασικό είναι ότι ο προπολογισμό θα καθορίσει το μέλλον της ΚΑΠ και το επίπεδο στήριξης που θα χορηγηθεί τελικά. Και θα είναι μια μακροσκελής και δύσκολη συζήτηση. Αλλά να ρωτήσω τα μέλη της Επιτροπής. Είπατε στην έκθεσή σας ότι υπάρχει ένα κοκτέιλ ζενιοκτώνων, αλλά δεν ε, μιλάτε για ε, την ανάπτυξη και εξέλιξη στην τεχνολογία που σίγουρα θα μας βοηθήσει να προοδεύσουμε. Στην παράγραφο 61 ζητάτε τη γνώμη μας για το ευρωπαϊκό ε, δίκαιο σε ό,τι αφορά συγκεκριμένους κλάδους και την επιστημική ασφάλεια. Εμείς σίγουρα θέλουμε να προωθήσουμε την τοπική παραγωγή, όμως ε, η Επιτροπή προτείνει αυτό να συμπεριληφθεί στο ευρωπαϊκό δίκαιο. Ευχαριστώ κύριε Πετήρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τα μέλη της Επιτροπής των Περιφερειών για τις προτάσεις τους. Νομίζω ότι αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή και πολύ επίκαιρη συζήτηση για το μέλλον της κοινή γεωρικής πολιτικής με την γεωργική πολιτική ώστε να καταστεί πιο αποτελεσματική. Ε, εντοπίσαμε τη μεγάλη αστάθεια των τιμών ε, στην αγορά, των προθεσμιών πληρωμής. Όλα αυτά ταλανίζουν τους γεωργούς. Θα πρέπει λοιπόν ε, να λάβουμε κάποια μέτρα για να τους βοηθήσουμε, γιατί τους ε, και να δίνουν απασχόληση σε ένα μεγάλο κλάδο γιατί 22 εκατομμύρια θέσει απασχόληση ε, ε, δημιουργούνται στη Γεωργία. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό κλάδο για ολόκληρη την οικονομία τη Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό φαίνεται και από τον προπολογισμό των γεωργικών. Λιγότερε διοικητικέ διατυπώσει και επίσης να έχουμε πιο δίκαιη, ακριβοδίκαιη κατανομή μεταξύ των επιχορηγήσεων, ώστε να ευνοηθούν από τις ενισχύσεις οι μικρές οικογενειακές βιορικές εκμεταλλεύσεις και όχι οι μεγάλες βιομηχανικές εκμεταλλεύσεις μόνο. Επίσης, να επιστήσουμε την προσοχή μας, ασφαλίσουν και να διαφυλάξουν τη δυναμικότητά τους και γι' αυτό χρειαζόμαστε αποτελεσματικά μέτρα για να βοηθήσουμε τους νέους αγρότες. Γιατί ε, και η απασχόληση των... Ο κύριος Κρόσο, εισηγητής. Είναι λίγο δύσκολο να συνοψίσω όλα όσα υπόθηκαν μέχρι τώρα, αλλά ίσως θα ήταν σκόπιμο να δώσω κάποιες απαντήσεις σχέση με κάποιες από τις τοποθετήσεις σας. Βεβαίως ε, και είναι λίγο δύσκολο να συνοψίσω όλα όσα υπόθηκαν μέχρι τώρα, αλλά ίσω θα ήταν σκόπιμο να δώσω κάποιες απαντήσεις σχέση με κάποιε από τι τοποθετήσεις σας. Βεβαίω ε, και των περιφερειών, η ΚΑΠ, θα πρέπει να τις ε, διαφυλάξει στο βαθμό Ας μην προχωρούμε λοιπόν με αυτοματισμούς προς την κατεύθυνση αυτή και επίσης το όραμα μια ΚΑΠ. Τίνει προς την αντίθετη κατεύθυνση. Και βεβαίως εδώ έχουμε και όλα τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την απασχόληση και όλες τις μεγάλες που νομίζω μας αποκαλύπτουν μια πραγματική πρόκληση. Όχι μόνο πόσο σημαντική είναι η προστασία του περιβάλλοντος και η σύνδεση χημικών προϊόντων, εκείνων δηλαδή που είναι ζημιογόνα για το περιβάλλον, και ταυτόχρονα αν αυτό στηριχθεί και από τις περιφέρειες, γιατί θα πρέπει οι περιφέρειες να έχουν σημαντικό ρόλο στην Ταυτόχρονα η έκθεση μας, έκθεση της Επιτροπής των Περιφερειών που έχουν ε, εγκρίνει στην πλειοψηφία τους τα μέλη μας, των ενώσεων, των συνδικαλιστικών, των ε, σωματείων και όπως υπόθηκε νωρίτερα και από τον κύριο Αντριού προτείνουμε σε και υπενθυμίζω εδώ ότι το τωρινό μοντέλο οδηγεί τοποθετήθηκαν να συνδυαστεί η γεωργία με την ανάπτυξη της υπαίθρου. Θα πρέπει δηλαδή μελλοντική ΚΑΠ να λάβει υπόψη. Περιβάλλον και υγεία και δημόσια υγεία. Εάν συνεχίσουμε, το ξαναλέω, στο μοντέλο που έχουμε αυτή τη στιγμή, δηλαδή μεγέθυνση διαρκής, γεωργικό κόσμο, ότι ανησυχεί όλο και περισσότερο για το μέλλον της γεωργίας, ιδιαίτερα εδώ στην Ευρώπη, στο διεθνές εμπόριο τώρα για να σταθμόριο και με παραγωγούς οι οποίοι δεν θα είναι σε θέση να διαθέσουν τα προϊόντα τους. Πολλά μπορούν να γίνουν οπωσδήποτε. Well, uh... Και ο πρόεδρος της Επιτροπής ΝΑΤ, ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για τις παρεμβάσεις σας και χαίρομαι που τα θέματα που πραγματευτήκαμε και εμείς στην έκθεση του κυρίου Κρός απασχολούν και εσάς. Υπάρχει απόλυτη σύμπτωση ως προς τη σημασία των θεμάτων και ελπίζω ότι η αγαστή μας συνεργασία θα συνεχιστεί και στο μέλλον και χαίρομαι που ο κύριος Σεκέρσκι συμμετείχε μέχρι στιγμή σε πολλές ε, εκδηλώσει και συνεδριάσει που οργανώσαμε στην Επιτροπή Περιφερειών και πιστεύω ότι και στο μέλλον θα δώσει το παρόν πάλι. Σας ευχαριστώ για το σχόλιο και για το χρόνο που και εμείς. Και σίγουρα το έργο δεν σταματά εδώ. Γιατί το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο ε, θα λάβουμε τότε στην Επιτροπή Γεωργίας την νομοθετική πρόταση και θα έχουμε κάτι πολύ πιο απτό για να σχολιάσουμε. Επίσης, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω γιατί εσείς ως ε, περιφέρειες και τοπική αυτοδιοίκηση είστε πολύ πιο κοντά και στο πλευρό των γεωργών και ε, πρώτα σε εσάς απευθύνονται οι γεωργοί για τα προβλήματά τους. Και πιστεύω ότι θα πρέπει και οι περιφέρειες και οι τοπικοί ε, να εντείνετε τις επαφές σας και με τους ευρωβουλευτές. Γιατί ε, είμαστε στις ίδιες εκλογικές περιφέρειες, ώστε καλό θα ήταν να έχουμε συνεργασία και να πείσουμε όλους για το επίπεδο χρηματοδότησης. Ε, έγινε αρκετές ε, προσδοκίες ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση και της ε, κοινή γεωργικής πολιτικής και της ε, πολιτικής συνοχής και μακάρι να επιβεβαιωθούν. Σας ευχαριστώ λοιπόν θερμά και πάλι για τη συμμετοχή και τη συνεργασία και να περάσουμε στο δεύτερο τμήμα της συζήτησης καλωσορίζοντας θερμότατα τα μέλη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της ΕΟΚΕ. Τα τρία που είναι ο εισηγητής για τον πιθανό μετασχηματισμό της κοινή διορικής πολιτικής, γνωμοδότηση του Ιουνίου του 2017. Επίσης έχουμε την κυρία Γιάρμιλα Ντουμπράφσκα από την ομάδα 1, τους εργοδότες. Ένας μας από την ΕΟΚΕ είναι ο κύριος Πέτερ Σμιτ από την ομάδα 2, τους εργαζομένους. Ε, ο κύριος Σμίτ είναι εισηγητής ε, στη γνωμοδότηση που αφορά τη συμβολή της κοινωνίας των πολιτών στην ανάπτυξη μιας σφαιρικής επισητιστικής, επισητιστικής πολιτικής. Ε, επίσης θα ήθελα να καλωσορίσω τον κύριο Μπρένταν Μπέρς που είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής ΝΑΤ, της Επιτροπής του Αντουμπραυσκά και τον κύριο Σμιτ που θα έχουν στη διάθεσή τους από τρία λεπτά ο καθένας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση που μας απευθύνατε προς την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Εκ την Ιρλανδία ε, έχω βοσκοτόπους και κατανοώ ιδιαίτερως ε, το πώς γνωριστεί στη συνθήκη τη ε, Ρώμη. Θεωρούμε ότι οποιαδήποτε επικαιροποίηση και αναμόρφωση της κοινή γεωργική πολιτική θα πρέπει να εξυπηρετεί τον στόχο της προστασίας του Ευρωπαϊκού 34 εκατομμύρια θέσει εργασία που εξαρτάται από τη γεωργία. Η ΕΟΚΕ στηρίζει την διατήρηση του συστήματος ανανέωση και επενδύσεις για τη στήριξη των ευάλωτων τομέων και περιοχών και ως ανάπτυξη του ΟΗΕ, ε, τους στόχους ε, υπό την COP21. Ε, για να αντιμετωπίσουμε τον θα πρέπει να βασιστούμε σε ένα πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο με προστασία του περιβάλλοντο με ότι τα, τα μέτρα της οικολογικής διάστασης του greening είναι πολύ περιοριστικά. Θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη-μέλη για την ε, προστασία της βιοποικιλότητας ε, των ε, υδροβιοτόπων και ούτω καθεξής. Αυτό θα βοηθήσει περισσότερους γεωργούς. Η ΟΚΕ προτείνει συνδεδεμένες πληρωμές για τις ευάλωτες περιοχές για να αποτρέψουμε την εγκατάλειψη της γης. Έχουμε σημαντικό πρόβλημα κατάληψη της γης σε όλη την Ευρώπη και στην Ιρλανδία και απαιτούνται συνδεδεμένε πληρωμές για να διατηρήσουμε τι καλλιέργειε. θα πρέπει να αυξηθεί ε, η παράδοση προϊόντων από τους ε, παραγωγούς και γεωργούς με την χρήση ε, των απλούστερων. Ο γεωργός λαμβάνει την επιδότηση την επόμενη χρονιά και αυτό είναι επιζήμιο για αυτούς. Ε, πρέπει να υπάρχει μέρημνα και ε, ένα πλαφόν για τον κάθε μονομένο ε, γεωργό και περαιτέρω σύγκληση μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Σε ό,τι αφορά τώρα και βιωσιμότητα δεν πρέπει να μπαίνουν στην ίδια πρόταση, δεν έχουν καμία σχέση. Να διασφαλίσουν λοιπόν ένα ίσο πεδίο ανταγωνισμού, σωστή ισορροπία για την προστασία της απασχόλησης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους ε, ευρωβουλευτές και να πω ότι νιώθω τιμή που βρίσκομαι εδώ σήμερα και μάλιστα ακόμη είμαστε όλους μας, αλλά πιστεύω ότι θα επιβιώσουμε και θα προετοιμάσουμε τις ε, και θα συνεχίσουμε να αξιο... εξαρτόμαστε από τη γεωργία. 7 εκατομμύρια γεωργοί και 7 εκατομμύρια γεωργικές εκμεταλλεύσεις παράγουν τρόφιμα. Δεν μας ενδιαφέρει το μέγεθος μιας γεωργικής εκμετάλλευσης. Γιατί, για παράδειγμα, 48% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων είναι μικρές οικογενειακές εκμεταλλεύσεις των αγροτικών γεών και λαμβάνουν το 22% των ενισχύσεων του γεωργικού προϋπολογισμού σε σχέση με το, με το 60% των μεγάλων. Θα πρέπει λοιπόν να εξασφαλίσουμε καλές συνθήκες για όλες τις εκμεταλλεύσεις, άσχετα του μεγέθους τους. Και όπως αναφέρεται και στην γνωμοδότηση, η ισότητα μεταξύ των κρατών μελών, μεταξύ των μεγάλων και των μικρών, μεταξύ των βόρειων και των νότιων κρατών, των ανατολικών και των δυτικών είναι σημαντική. Και να μην ξεχνούμε, είναι σημαντική και η ισότητα μεταξύ των νέων αγροτών και των πιο ηλικιωμένων αγροτών. Θα πρέπει αυτή την ε, ισότητα και τη δικαιοσύνη μεταξύ όλων αυτών. Η αλήθεια είναι ότι μία και μόνο πολιτική δεν είναι θαυματουργή και δεν μπορεί να λύσει όλα τα προβλήματα. Η κοινή γεωργική πολιτική είναι μία μόνο από τις κοινοτικές πολιτικές. Κάθε πολιτική όμως στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχει και μία γεωργική διάσταση, να συνδέεται με τη γεωργία. Είναι ώστε το τοπίο που θα διαμορφωθεί να είναι όμορφο. Σας ευχαριστώ και ελπίζω ότι η αναθεωρημένη κοινή γεωργική πολιτική, η αναμορφωμένη ΚΑΠ θα δημιουργήσει ένα ωραίο εργασιακό χώρο και για όλους μας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να εκφράσω τις ευχαριστίες μου και για την πρόσκληση και για τη δυνατότητα να τοποθετηθούμε εδώ και να προβούμε σε ανταλλαγή απόψεων μας. είμαι Πρόεδρος της μόνιμης ομάδας μελετών για βιώσιμα συστήματα παραγωγής στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στόχος μου είναι να σας παρουσιάσω το ζήτημα της βιωσιμότητας σε σχέση με τη Γεωργία. Η κατάσταση λοιπόν που περιγράφηκε αρκετές φορές σήμερα ήταν ότι δεν χρειάζεται να εφεύρουμε τα πάντα, αλλά ότι έχουμε μια κατάσταση στο σύστημα παραγωγής των τροφίμων που δεν λειτουργεί απόλυτα ικανοποιητικά. Πρέπει λοιπόν να διαρωτηθούμε πρώτα απ' όλα, έχουμε όντως σύστημα παραγωγής τροφίμων. τροφίμων. Ναι, υπάρχει, αλλά δεν είναι ενιαίο δεν καλύπτει τους πάντες. Υπάρχουν συστήματα παραγωγής τροφίμων στην Ευρώπη τα οποία ε, αναπτύσσονται από διάφορους φορείς, πρωταγωνιστές εμπλεκόμενους που όμως δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι δηλαδή συστήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενώ υπάρχει μια κοινή γεωρική πολιτική δεν ε, υπάρχει αυτή η γενική θεώρηση και πολλοί είπαν σήμερα ότι κάτι τέτοιο είναι αυτό που χρειαζόμαστε. Υπόθηκε από πολλού ομιλητέ ότι είναι κατακαιρματισμένη η εικόνα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρουσιάστηκε και νωρίτερα άλλωστε ε, μια έκθεση, τη οποία εγώ είχα αναλάβει την ε, διατύπωση, με 5-6 ε, γενικέ διευθύνσει παρούσε που είχαν να πούνε πράγματα για την αγορά των τροφίμων. Κατακαιρματισμένη λοιπόν η εικόνα της ε, παραγωγής και αγορά τροφίμων ε, και πρώτη μας διαπίστωση ότι χρειάζεται μια ενιαία προσέγγιση που να περιλαμβάνει τα εξής. Ας ε, περιγράψω την εικόνα ενός ναού. Ένας ναός ο οποίο θα έχει σαν στέγη μια ενιαία πολιτική και θα στηρίζεται πάνω σε διαφορετικούς πυλώνες πυλώνες οι οποίοι βεβαίως θα είναι μια κοινή γεωργική πολιτική Βεβαίως θα είναι ε, η, εδαφική, η ανάπτυξη της υπαίθρου, βεβαίως θα είναι και η βίωσιμη ε, παραγωγή και επεξεργασία τροφίμων, βεβαίως θα είναι και το ζήτημα, ο δημογραφικό στην ε, Γεωργία, η προστασία του περιβάλλοντος, εκπαίδευση, το, το εμπόριο, οι μεταφορές, όλοι αυτοί οι πυλώνες λοιπόν στηρίζουν τον ε, ναό αυτών που παρουσιάζεται τέτοια πολυμορφία και πρέπει να, στηριχθεί, να στηριχθούν όλοι αυτοί οι πυλώνες σε, μία, ε, σε ένα θεμέλιο, σε μία βάση, σε ένα βάθρο. Εθνικά κράτη, αν αυτό συνεχιστεί θα έχουμε 28 διαφορετικά συστήματα σήμανσης τροφίμων. Ήδη στη Γαλλία έχει ξεκινήσει η αγωγή ενός συστήματος που όμως δεν τα οποία έχει, έχουν κηρύξει τη δεκαετία της διατροφικής ασφάλειας, ε, της επιστηστικής ασφάλειας. Έχουμε στόχους βιωσιμότητας των ΗΠΑ, τα οποία έχει, έχουν κηρύξει τη δεκαετία της διατροφικής ασφάλειας, ε, της επιστηστικής ασφάλειας. Έχουμε στόχους βιωσιμότητας των των Βρυξελών. Μια σειρά από πρωτοβουλίε λοιπόν και προσεγγίσεις που έχουν να κάνουν με τα τρόφιμα και τη γεωργική παραγωγή τροφίμων και που μας υποχρεώνουν και εμείς να στραφούμε στον τροφίμων. Γιατί πρέπει να είναι διαρκώς μειούμενες οι τιμές. Χρειαζόμαστε υψηλότερες τιμές στο χώρο των τροφίμων και η FAO έκανε πρόσφατα μία ψία της τροφής. Και αυτό έχει να κάνει με μία γενικότερη πολιτική για τα τρόφιμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι του καταναλωτή Εύνα. Σας ευχαριστώ. Και καλημέρα σας. Ε, δεν πρόκειται να καλύψω ζητήματα που επισήμαναν οι εμπειρογνώμονες μας. Θα αναφερθώ σε κάποια σχόλια των Ευρωβουλευτών που ε, αναφέρονται σε θεμελιώδη στοιχεία και την πραγματικότητα της υπαίθρου. Και εγώ έχω επιχείρηση σε μια τέτοια αγροτική απομονωμένη ζώνη και ξέρω πως ε, η κοινή πολιτική λειτουργεί στις αγροτικές αυτές περιοχές, τις απομονωμένες. Φυσικά μας ενδιαφέρουν ποιοτικά τρόφιμα από βιώσιμες πηγές, αλλά μέχρι στιγμής είναι πολύ φθηνά αυτά τα τρόφιμα. Είναι αποτρόπαινο Αυτό δεν το δέχονται και τόσο χαμηλές τιμές δεν μπορούν να τις δεχτούν οι νέοι. Γι' αυτό δεν έχουμε νέους στην Ήπεθρο. Θα σας πω τι μου είπε ε, ένας νέος ε, απόφυτος μετά από μια συνεδρία σε ΟΚΕ. Ένας από, πτυχιούχος ε, και η κυρία αυτή. Όχι. Γιατί ε, να πάω σε μια απομονωμένη αγροτική, αγροτική περιοχή, να είμαι οικονομικά και κοινωνικά σε δυσμενή θέση. Προς Τι Τι να της πω. έχει δίκιο. Η ευρυζωνικότητα δεν είναι να φτάνει μέχρι την υπεθρο. Η συγκίνηση. Οπότε το ζήτημα που ανακύπτει και το ερώτημα που ανακύπτει επανειλημμένως είναι τι θα κάνουμε για το εργατικό μας δυναμικό. Μία από τις επιχειρήσεις που έχω αφορά τη δασοκομεία. Ε, έχει άμεση σχέση ε, με την ΚΑΠ και με τη σπορά. Οι μηχανές, ε, ενώ είναι πολλές οι μικρές επιχειρήσεις που ασχολούνται με την υλοτομία και που δίνουν θέσεις απασχόλησης, αλλά δεν έχουμε εργατικό δυναμικό. Το εργατικό δυναμικό συγκεντρώνεται στα αστικά κέντρα. Και φυσικά έχουμε μεγαλύτερη ένταση γεωργίας λόγω των καλύτερων μηχανημάτων, αλλά σε μια θέση και να λειτουργούν τις μηχανές, να τις χειρίζονται. Κάποιος θα πρέπει να χειρίζεται αυτά τα μηχανήματα. Και οι θέσεις απασχόλησης ε, που θα χαθούν δεν θα είναι στη, στις αγροτικές περιοχές, αλλά και στα αστικά κέντρα. Υπάρχει ένα, ένα κόστο παντού στην Ευρώπη. Οπότε το ερώτημα παραμένει τι ενδιαφέρονται οι θύνοντες για τις απομονωμένες αγροτικές περιοχές. Γιατί αναφερθήκαμε στην επαγγελματική κατάρτιση και την εκπαίδευση. Ένας αρχιτέκτονας μου είπε εγώ δεν μπορώ να προσλάβω μαθητευόμενο, ασκούμενο, γιατί ο ασκούμενος θα πρέπει να πάει στο σχολείο του για μία μέρα και για να πάει στο σχολείο θέλει μισή μέρα για να δέσει υποδομές ώστε η επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση να γίνεται στις αγροτικές περιοχές. Και η ΚΑΠ είναι έτοιμη αυτή τη διαδικασία. Στα ζητήματα όμως είναι πολύ ευρύτερα. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε όλοι ότι μπορεί ε, η ΚΑΠ να είναι το ορατό τμήμα, αλλά είναι πολύ πιο ευρύες. Σας ευχαριστώ. Θα περάσουμε τώρα στη συζήτηση με τα μέλη της Επιτολόγου. Μπορεί να κλέψω τα λόγια του από το στόμα του κυρίου Φλάναγκαν και να πω πόσο λίγοι θα είναι, είναι σήμερα εδώ βουλευράς κοινοβουλίου για να συστηματική στήριξη για έναν γεωργό και τις ε, προσδοκίες για την ε, περιβαλλοντική στήριξη ότι είναι πολύ μεγάλη κλιματική αλλαγή, ότι φταίνει η γεωργία, άρα αυτοί θα πρέπει να αναλάβουν ε, και την αποκατάσταση. Εγώ για παρνά περιορίζω τι εκπομπέ οξυδίων του άνθρακα. Τι κάνω, χρησιμοποιώ λιγότερο τα τρακτέρ μου, περιορίζω την γεωργική μου λοιπόν δραστηριότητα ή πλέον δεν κόβω τα δέντρα μου για ε, να τα κάψω που έκανα πάντα. ή για παράδειγμα να έχω λιγότερα πρόβατα για να μην έχουμε εκπομπές και άλλες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Τι κάνω, σπέρνω λιγότερα ε, όσπρια. Πώς ε, περιορίζω και μετριάζω το όζον, κανείς δεν ξέρει. Αλλά όλα αυτά σημαίνουν ότι τελικά δεν θα έχω κανένα εισόδημα. Τις έχετε σκεφτεί όλες αυτές τις ανοησίες. Ο κύριος έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και ε, συμμερίζομαι τις απόψεις με τον, του προηγούμενου μιλητή. Είναι κρίμα που τόσο καλά αμοιβόμενοι ε, ευρωβουλευτές δεν μπορούν να έρθουν εδώ στη σημερινή συζήτηση και η μεγάλη ηρωνία είναι ότι έρχονται οι ευρωσκεπτικιστές να συζητήσουν το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώ οι άλλοι που είναι υπέρμαχοι δεν έρχονται. Πραγματικά είναι μεγάλη ηρωνία. Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων στη τελευταία κοινή γεωργική πολιτική, προφανώς και υπήρξαν συζητήσεις σε όλη την Ιρλανδία, αλλά και ευρύτερα πολλοί στις ε, μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και στις μειονεκτούς περιοχές. Ε, τους, λέγαμε, τους λέγανε μάλλον να περιμένετε τον ε, δεύτερο πυλώνα. Ε, αλλά τελικά δεν υπήρχε τίποτα. Παρότι μπορεί κάποιοι να λέγανε κάλιο πέντε και στο χέρι παραδέκα και καρτέρι, τελικά τίποτα δεν βγήκε από όλο αυτό. Και όταν έχουμε ένα κέικ, όταν κάποιος παίρνει τα πέντε κομμάτια του κέικ, οι υπόλοιποι προφανώ και θα μείνουν χωρί τίποτα. Αν όμω ε, η απόφαση για το ποιο θα πάρει περισσότερα κομμάτια λαμβάνεται από αυτόν που έτσι κι πάντα παίρνει μεγαλύτερο κομμάτι, τότε αυτό πρέπει να μας οδηγήσει σε προβληματισμό. Για τη νέα λοιπόν ΚΑΠ θα πρέπει ε, να δώσουμε ένα πλαφόν ε, εγώ προτείνω 20.000 ευρώ. Ε, κάποιοι λένε ότι αυτά είναι πολλά χρήματα, αλλά για αυτούς που παίρνουν 1.000, 2.000, 3.000 ευρώ, αυτό θα είναι πραγματικά σωτηρία και θα τους ε, κρατήσει στη γεωργία. Όπως ε, όταν έχουμε ένα σκύλο ξέρουμε ότι πρέπει να παρεμβούμε για να του δώσουμε τη σωστή ποσότητα τροφής, αλλιώς θα φάνε μέχρι θανάτου. Το ερώτημα λοιπόν που έχω εγώ και προς τον κύριο Μπραν συγκεκριμένα είναι στις επόμενες διαπραγματεύσεις πώς μπορεί κάποιο σαν και εσάς ε, να είναι αμερόληπτος ε, διαπραγματευτής για τους γεωργού όταν εσείς το 2016 λάβατε 55.000 ευρώ και δεν θα υπάρχουν τόσα χρήματα για όλους ε, στο μέλλον. Οπότε, πώς μπορεί κανείς να, να διαπραγματευτεί τη νέα ΚΑΠ ε, κάποιος που έτσι κι λαμβάνει τη μερίδα του λέοντος ε, από τα κονδύλια της ΚΑΠ και πώς θα είμαστε σίγουροι ότι εσείς θα τα κατανείμετε σωστά. Ρωτήστε και τους κατοίκους του Λίτρων που χάσαν 11 εκατομμύρια ευρώ την προηγούμενη περίοδο. Ε, θα κάνετε τα ίδια ε, με βάση ε, αυτά που γίνονται σήμερα. Πώς θα αλλάξετε αυτή την κατάσταση. Ο κύριος Ροπέ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τα μέλη της ΕΟΚΕ που ήρθαν στην Επιτροπή μας και μας παρουσίασαν τις γνωμοδοτήσεις τους. Όπως ακούσαμε και προηγουμένως, οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και οι δικές μας δεν συμπίπτουν πάντα. Θα ήθελα να σχολιάσω μερικά από τα σημεία των γνωμοδοτήσεών σας. Αναφέρθηκε επανειλημμένως ότι η ευρυζωνικότητα δεν είχαμε παρόλα αυτά βελτίωση των κοινωνικών συνθήκων. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το εισοδηματικό κενό, το εισοδηματικό χάσμα που υπάρχει μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών. Και για να γεφυρωθεί αυτό το χρηματοδοτικό και οικονομικό κόσμο στην Ήπεθρο, αλλά ούτε και αυτό θα λύσει το πρόβλημα. Θα πρέπει ο κόσμος όχι μόνο να επιστρέψει στην Ήπεθρο, αλλά και να παραμείνει εκεί. Και γι' αυτό θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ένα αξιοπρεπές εισόδημα ε, για να μπορεί κανείς να δουλεύει στην Ορβηγία αντί στην πατρίδα του. Στο παρελθόν είχαμε το σιδηρούν παραπέτασμα που εμπόδιζε τις μετακινήσεις, αλλά τώρα υπάρχει ένα νοητό παραπέτασμα εξαιτίας της ανισότητα που υπάρχει. Θα πρέπει για να καταπολεμηθεί αυτή η ανισότητα να έχουμε μια πιο ακριβωδική κατανομή του γεωρικού εισοδήματος και αυτό θα πρέπει να λάβουμε υπόψη στην επόμενη αναθεώρηση της ΚΑΠ. Σε ό,τι αφορά τις τιμές των τροφίμων, συμφωνώ ότι θα μπορούσαμε να έχουμε και ακριβότερα τρόφιμα. Δεν του εισοδήματο στην αλυσίδα τροφίμων. Αν αυτή η ισότητα δεν αποκατασταθεί, το πρόβλημα θα εξακολουθεί να ισχύει. φόρους ε, για τα τρόφιμα, αλλά δεν καρπώνεται τα εισοδήματα αυτά ο παραγωγός, ο κύριος Νίκολσον. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ τον κύριο Μπρέν για τα σχόλιά του και για τη δουλειά Η κατάσταση θα είναι πάρα πολύ δύσκολη για τους γεωργούς και κτηνοτρόφους και για το 20. η κατάσταση θα είναι πάρα πολύ δύσκολη για τους γεωργούς και εκτινοτρόφους και για 28 και για 27 κράτη-μέλη. Δεν πρέπει να το λησμονούμε αυτό, σας διαβεβαιώ. Για τα σχόλια του κυρίου Άγνου και άλλων σε σχέση και το υπεγράμμισε ο κύριος θα υπάρχουν ε, κενά 12 δισεκατομμυρίων, ε, εκ των οποίων προτείνεται τα 6 δισεκατομμύρια να προκύψουν από εξ... Ο Θεός να μας φυλάει, θα εξαρτώμαστε από τον κύριο Γκόβαν για τα θέματα που αφορούν την γεωργία και την επιβίωση των γεωργών μας. Τέλος πάντων, άλλα είναι αυτά τα προβλήματα της γεωργίας ή της παραγωγής τροφίμων. Καμία εθνική κυβέρνηση, κανένας επίτροπος ή Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είχε τη διάθεση αλλά και την Παρισία να αναλάβει σχετική παρουσία, Παρισία, είτε πρόκειται για τη Σκωτία, είτε για τη Γερμανία, την Ιταλία ή οτιδήποτε άλλη γωνιά της Ευρώπης, δεν πρόκειται να αλλάξει αυτό. Έχει φτάσει η κατάσταση σε κάποιους που είναι ιδιαίτερα ισχυροί, που υπαγορεύουν ε, τη διαμόρφωση των τιμών και την κατάσταση των προϊόντων και έτσι ο νέος γεωργός και τις μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες τον πληρώνουν, τον ενισχύουν στην αρχή αλλά στη συνέχεια είναι δεσμευμένος σε φόρους ζωής να τους ξεπληρώνει τα χρεωστούμενα. Ε, πολλά στον κόπο και το μόχθο. Ε, και έτσι σε 10-20 χρόνια θα πρέπει να γίνουν πιο αυστηρά τα τρόφιμα, μοιραία θα γίνουν πιο, αυστηρά, πιο ακριβά τα τρόφιμα γιατί δεν θα υπάρχουν τόσοι γεωργοί. Ευχαριστώ κύριο Σβάιτς. Στα αγγλικά πολλά υπόθηκαν, πολλά από τα σημαντικά και θέλω να ευχαριστώ τον Τζον Μπράιν, εισηγητή για το εξαιρετικό του έγγραφο. Ένα πολύ σημαντικό θέμα ε, μοντέλο γεωργίας αναφέρεται, αναφέρεστε σε ε, γεωργικούς συνεταιρισμούς, οικογενειακές εκμεταλλεύσεις και εταιρείε γεωργικές. Τι εννοείται με τον όρο εταιρείες που μπορεί να φέρει καλά αποτελέσματα χωρίς ζημιά στο περιβάλλον ε, όπως γίνεται τώρα, όπως ε, υπάρχει ζημιά. Υπάρχει ω προ αυτό. Για ε, εκείνον που είναι προ τα αριστερά μου, κάποιο ο οποίο μπορεί να εισπράττει 50.000 ευρώ το χρόνο, εάν κάνει δουλειά καλή, αν έχει γεωργική παραγωγή, αν προσφέρει ε, ο παραγωγό ο οποίο θα εισπράξει 30-40.000 ή 50.000 βεβαίως εφόσον κάνει σωστά τη δουλειά του ω ε, γεωργική εκμετάλλευση. Και τελευταία λόγια, η ΚΑΠ πρέπει να μιλούμε επομένω, όχι για λύσει ε, παροχής διατροφική ασφάλεια. Πολύ ευχαρίστω να έρθω να ρίξω μια ματιά στη δική σα γεωργική εκμετάλλευση. Δεν ξέρω το όνομά σα. Και ελάτε κι εσεί να ρίξετε μια ματιά στη δική μου φάρμα. Η περισσότερη γεωργία που ασκώ δεν ε, λαμβάνει επιδοτήσεις. Είναι παραγωγή ε, αυγών από κοτόπουλα ελευθέρας βοσκής. Και αν θέλετε να με... Δεν τα δίνετε καλύτερα κανένα ραντεβού να πιείτε ένα καφέ μαζί και να ανταλλάξετε απόψη για να μην συνεχίζουμε τη συζήτηση. Ε, θα επανέλθω σε αυτό το θέμα. Α, δώσατε σε άλλον το λόγο. Δεν πρέπει να γίνεται συζήτηση επί προσωπικού. Ας α, επικεντρωθούμε σε ευρύτερα ζητήματα, όχι σε προσωπικά. Ο συνάδελφος Φλάναγκαν έχει δίκιο ότι οι παρόντες στην αίθουσα είναι περισσότερο ευρωσκεπτικιστές αλλά είμαστε έχουμε έναν βιώσιμο γεωρικό προϋπολογισμό και μετά το Brexit αυτό θα είναι πολύ δύσκολο να διαφυλαχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μερικά αυτά ζητήματα, μερικοί, όπως ο κύριο Άγνιο, βλέπουν προβλήματα. Εγώ όμως πιστεύω ότι μπορούμε να βρούμε τρόπους για να τα συμφιλιώσουμε και να έχουμε μια παραγωγή που θα έρθει και ακόμη για τη μελλοντική χρηματοδότηση της γεωργίας και για την στήριξη των ενεργών και παραγωγικών γεωργών θα πρέπει να εξετάσουμε το θέμα και της επισητιστικής ασφάλειας. Πιστεύω ότι θα πρέπει να είμαστε πιο συνεπείς και πιο συνεκτικοί στις χρηματοδοτήσεις μας. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα για την αγροτική ανάπτυξη από το δεύτερο πυλώνα της ΚΑΠ θα πει των διαρθρωτικών ταμείων, του Ταμείου Συνοχή και των χρηματοδοτήσεων του δεύτερου πυλώνα. Κύριε Ντελαέ. Προπολογισμό τη κοινή γεωργική πολιτική. Θα ήθελα όμω να επισημάνω και να υπενθυμίσω αυτό που ανέφερε ο πρόεδρο Γιούγκερ πρόσφατα. Είπε ότι τα κράτη-μέλη που θεωρούν ότι αρκεί να μειώσουν τι ε, ε δαπάνε με το περιβάλλον. Δεν ισχύει όμω αυτό. Θα πρέπει στην επόμενη κοινή γεωργική πολιτική να το εξετάσουμε προκειμένου. Μάλιστα, έχετε δίκιο. Σίγουρα θα είναι σημαντικό πρόβλημα ε, το Brexit και ο προπολογισμό. Ακούσαμε τον Επίτροπο Έτιγκερ να λέει ότι θα υπάρχει ζήτημα και είναι και θέμα με τη διαμόρφωση κυβέρνηση τη ε, του περιβάλλοντος. Στην τελευταία διαφάνεια που είδατε ανέφερε και τα προγράμματα χαμηλών εκπομπών. Ξέρουμε ότι είναι πιο δαπανηρές, αλλά έτσι γίνεται. Δεν ε, γίνεται να τα κάνουμε όλα με πολύ χαμηλό κόστος σε οικολογικές καταστροφές, ψήλους των δασών και το καθεξής. Οπότε δεν έχει κανένα νόημα όλο αυτό εμείς ε, να παράξουμε τροφή με βιώσιμο τρόπο. Αν δείτε την Κίνα, 20% του παγκόσμιου πληθυσμού, περίπου 7% της γης και μειώσει το περιβάλλον. Υπάρχουν λοιπόν τέτοιες προκλήσεις. Ε, όταν αυξηθεί ο πληθυσμός του πλανήτη στα 9 ή και στα 11 δις, ε, αυτό θα έχει νέο αντίκτυπο. Η νέη γεωργοί, τεράστια πρόκληση και αυτή. πολύ το ανέφερα σήμερα το πρωί. Το θέμα είναι το εισόδημα και παίρνουμε το 1 τρίτο του μισθού που παίρνει ο κύριος Φλάνναγκαν ε, που είναι εδώ. Είπατε το 20.000. Κανένα πρόβλημα δεν θα είχα με αυτό το εισόδημα. Αλλά αυτή δεν είναι μόνο η δική μου γνώμη. Είναι η γνώμη των ε, σωματείων, των εργοδοτών, των καταναλωτών της κοινωνίας των πολιτών. Έγινε μεγάλη συζήτηση και εμείς πιστεύουμε στην ε, περαιτέρω αναδιανομή να τεθεί πραγματικά ένα πλαφόν Κάποιοι πρότειναν τα 100.000, άλλοι λιγότεροι, αλλά είναι δύσκολο να θέσουμε έτσι ένα, ε, μία τιμή, γιατί εξαρτάται και από τη χώρα. Εγώ πραγματικά πιστεύω στην ε, οικογενειακή γεωργία, αλλά είναι διαφορετικό το μοντέλο στην Ανατολική Ευρώπη. Στις διαπραγματεύσεις ε, μιλήσαμε για τους συνεταιρισμού, αλλά και επιχειρήσεις που υπάρχουν στην Ανατολική Ευρώπη. Είναι πιο περίπλοκα λοιπόν τα πράγματα. Ε, προτάθηκε το 100.000 ευρώ, καμία σχέση με το 1 εκατομμύριο που λέγατε εσείς προηγουμένως. Αλλά η, η παράδοση των γεωργικών προϊόντων είναι το πιο σημαντικό. Ε, υπάρχει σημαντικό κόστος. Συχνά αναφέρεται το παράδειγμα της Νέα Ζηλανδία που έχει καταργήσει εδώ και 20 χρόνια τις επιδοτήσει. Αλλά αναπτύχθηκαν οι μεγάλες επιχειρήσεις των ζώων. Πρέπει λοιπόν εμείς να προσπαθήσουμε να προστατεύσουμε το ευρωπαϊκό μοντέλο οικογενειακής γεωργίας. Αυτό θα βοηθήσει και τους νέους γεωργούς. Γιατί πρέπει να διασφαλίσουμε και την πρόσβαση των νέων και στις επιδοτήσεις. Σαφώς και απαιτείται περαιτέρω σύγκληση.